Uh, good afternoon. Um, Η πρόεδρος κυρία Άννα Γκόμες. Καλώς ορίσατε μέλη της Επιτροπής καθώς και μέλη που παρίστατε ως ακροατήριο για να συζητήσουμε πρόκειται για την τελευταία συνεδρία σε ό,τι αφορά το πανεπιστημιακό fact-finding. Είχαμε κάνει παρόμοια συνεδρίαση και τον Απρίλιο, στις 27 Απριλίου. Και τα σχετικά απορίσματα ανεβρίσκονται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Είναι αυτονόητο ότι οι μελέτες που παρουσιάζονται είναι αναπόσπαστο μέρος της πορείας των εργασιών μας. Σήμερα θα ε, παρουσιαστούν τρεις μελέτες που χωρίζονται σε δύο ξεχωριστά πάνελ. Το πρώτο αναφέρεται στον ρόλο που παίζουν διαμεσολαβητές, δικηγόροι, τραπεζικοί κλπ. και στους κανόνες που ε, εφαρμόζονται στα πρόσωπα αυτά. Το δεύτερο πάνελ αναφέρεται στις πρακτικές offshore σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και υπερπόνητες κτήσεις εδάφη, ιδίω της Γαλλίας, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και των κάτω χωρών. Δυστυχώς και ε, λόγω αλλαγή της τελευταία στιγμή στην ημερήσια, μάλλον στην, ε, στην, ε, στις του Υπουργού Εξωτερικών του Εκουαδόρου κ. Λόγκ, δεν θα μπορέσει ο ίδιο να είναι παρόν σήμερα. Θα προχωρήσουμε αμέσω λοιπόν και θα ήθελα να εξηγήσω ότι η παρουσίαση των δύο μελετών στο πρώτο πάνελ θα καταναλώσει 25 λεπτά η κάθε μία και για το δεύτερο πάνελ έχουμε τρεις ομιλητές στους οποίους θα διαθέσουμε το 15 λεπτά κατά το μέγιστον. Μετά από κάθε πάνελ θα διεξαχθεί γύρω συζητήσεων, ερωτήσεων και απαντήσεων με τα μέλη της Επιτροπής. Θα ε, τίθενται ερωτήσεις για διαστήματα 5 λεπτών, δηλαδή ένα λεπτό για την ερώτηση και το υπόλοιπο για την απάντηση. Εάν το επιτρέψει ο χρόνος, τα μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν και δεύτερη ερώτηση, χωρίς όμως να υπερβούν το όριο των πέντε λεπτών. Έχοντας υπόψη ότι δεν έχουμε και έγγραφα με την ε, μορφή του χαρτιού, διότι ε, ε, λειτουργεί το κοινοβούλιο όσο γνωρίζετε τώρα χωρίς έγγραφα, δηλαδή paperless. Μπορείτε όμως να βρείτε όλα τα στοιχεία που θέλετε στην ιστοσελίδα της ε, Επιτροπής, της Εξεταστικής μας Επιτροπής. Και βεβαίως αναμεταδίδεται από το διαδίκτυο η συζήτησή μας. Έχετε υπόψη σας ότι κάθε φορά που κάποιος ομιλητής ε, πατά το κουμπί του μικροφόνου του, η κάμερα ε, δείχνει το πρόσωπό του. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στο πρώτο πάνελ που αναφέρεται στον ρόλο των διαμεσολαβητών και στους κανόνες που διέπουν τα των δραστηριοτήτων τους και θα παρακαλέσω τον κύριο Πέτερ Τεγκρούν που είναι ερευνητής Research Fellow στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών, ΣΕΠΣ. Τον παρακαλώ λοιπόν να λάβει το λόγο για να παρουσιάσει την μελέτη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πριν αρχίσω την παρουσίασή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή Πάνα καθώς και την Γραμματεία που μας επέτρεψε να μελετήσουμε τον ρόλο των διαμεσολαβητών στην, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της ε, Επιτροπής Εξετάσεως των Εγγράφων Παναμά. Θα αρχίσω με τα βασικά στοιχεία των Εγγράφων Παναμά που έχουν ε, σημασία για τη σημερινή συζήτηση για τον ρόλο των διαμεσολαβητών. Μετά θα περάσω στον κύκλο λήψεως των αποφάσεων. Πρώτα θα παρουσιαστεί ο ρόλος των διαφόρων φορέων και μετά θα προχωρήσω στην συζήτηση των επιμέρους φορέων. Θα ολοκληρώσω με μερικές συστάσεις που έχουν τον στόχο να ενθαρρύνουν την λήψη δράσης. Σε ό,τι αφορά τα έγγραφα Παναμά, για να δείξω ας πούμε έναν ισταντανέ πραγμάτων που έχετε ήδη δει προηγουμένως, αλλά είναι και σημαντικό να κατανοήσουμε τα πορίσματα της μελέτης μας, περίπου 214.000 νομικά πρόσωπα offshore, υπεράκτια. Αν θα είδατε ότι μόνο το 1 τέταρτο περίπου από αυτά, δηλαδή 55-56 περίπου εξακολουθούν να είναι ενεργά από τους φορείς αυτούς, ο αριθμός των ενεργών αυτών οντοτήτων αυξανόταν μέχρι το 2008 και μετά να μειώνεται. Και το 2013 είδαμε από τότε να μειώνεται ο αριθμός των ε, νομικών αυτών προσώπων υπεράκτιας δραστηριότητας. Το ερώτημα είναι αν έχουν μειωθεί και οι δραστηριότητές τους. Υπάρχουν κάποιοι υπολογισμοί που δείχνουν ότι συνεχίζει να αυξάνεται η δραστηριότητα αυτή. Φαίνεται πως πάντως εμπλέκονται σε αυτές λιγότερες οντότητες. Και εξετάζοντας αυτές τις οντότητες βλέπετε ότι η Μοσακ Φονσεκά δραστηριοποιούνταν στις ε, Σεϊχέλες, στο Βρετανικό, ε, Βρετανικές υπερπόδειε κτίσεις κλπ. δεν ε, υπάρχει πλήρης επισκόπηση όλων των υπερπόντιων αυτών δραστηριοτήτων. Η μελέτη μας εξέτασε τα έγγραφα Παναμά που ανέρχονται στο 5 10% των, των συνολικών δομών offshore. Ο ρόλος των διαφόρων συμβούλων και διαμεσολαβητών βλέπετε, αν βλέπετε τώρα στην οθόνη το γράφημα, βλέπουμε λοιπόν ότι Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ομάδες ε, δρόντων προσώπων, ας το, πω, ας το έτσι. Υπάρχουν πρώτα αυτοί οι οποίοι δίνουν τις συμβουλές για την δημιουργία των υπερπόνδιων δομών. Μπορούν να είναι πλούσια άτομα, μπορούν να είναι και εταιρείε. Συνήθως είναι εύπορα πρόσωπα. Το βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί σήμερα είναι η σύμβουλοι και ενδιάμεση. Βλέπετε συχνά ότι δεν λειτουργούν μόνοι τους, αλλά σε συνδυασμό μεταξύ τους και μπορεί να έχουν διαφορετικές δομές. Στο γράφημα προσπαθούμε να απλουστεύσουμε με κατανοητό τρόπο το πώς λειτουργούν, αλλά ταυτόχρονα να δώσουμε και με αφαιρετικό τρόπο. Βλέπετε στην τρίτη ομάδα διαμεσολαβητών είναι πρόσωπα που είναι οι δημόσιες αρχές που έχουν και εκεί διαφορετικούς ρόλους αφενός, δηλαδή υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι αρμόδιο, μπορεί να συμμετέχει αλλά μπορεί και όχι ως δημοσιονομική αρχή η οποία μπορεί να παίζει και εποπτικό ρόλο εποπτικό ρόλο επί των συμβούλων και διαμεσολαβητών. Και εδώ λοιπόν οι ε, δημοσιονομικές αρχές είναι αρμόδιες και για την επιβολή των νομοθετικών διατάξεων. Έρχομαι τώρα σύντομα στον ρόλο των διαφόρων αυτών μερών και θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τέσσερα ερωτήματα σχετικά με κάθε μια από τις ομάδες αυτής. Ποιος κάνει τι, πού. Διότι σημαντικό είναι όχι μόνο το τι κάνουν τα άτομα αυτά, τι κάνουν, είναι σύμβουλοι, είναι διαμεσολαβητές, τι είδους διαμεσολαβητές ή ενδιάμεση και πού διεξάγονται οι δραστηριότητε αυτέ, γιατί θα δούμε ότι οι περισσότερε από αυτέ τι δραστηριότητε λαμβάνουν χώρα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα είναι δύσκολο λοιπόν για ε, εσά εδώ να νομοθετήσετε. Ίσως χρειαστεί λοιπόν να ψάξετε να βρείτε άλλε λύσει και να συνεργαστείτε με άλλου φορεί. Θα δούμε επίση ότι υπάρχουν πολλών ειδών σύμβουλοι και ενδιάμεση σε διάφορα στάδια της δημιουργίας και διατήρησης και χορήγηση συμβουλών στις διάφορες δομές. Πόσο σημαντικοί λοιπόν είναι οι σύμβουλοι και οι διαμεσολαβητές στις δομές αυτές. Και πολύ σημαντικό είναι επίσης όταν θα φτάσουμε στην τελική φάση πλέον ε, της μελέτης, πολύ σημαντικές εκείνοι οι συστάσεις. Ας δούμε λοιπόν τώρα τους ε, απότερους ε, πραγματικούς κυρίους. Θα δούμε στα δεδομένα αυτών των πολλών χιλιάδων ε, δομών και θα δούμε σε αυτές που είναι ε, ακόμη δραστήριες και που είναι περίπου 56.000 από αυτές τις offshore, ψάξαμε να βρούμε ποιοι κρύβονται από πίσω. Εξετάζοντας τα δεδομένα των μετόχων, είδαμε, όταν τα εξετάσαμε αυτά, ε, είδαμε αμέσως ότι για πολλές από τις δομές αυτές, παρόλο που έχουν αποκαλυφθεί τα έγγραφα αυτά, δεν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε ποια είναι τα πραγματικά πρόσωπα που κρύβονται από πίσω. Για το 25 περίπου της 100 των ε, δομών αυτών, αυτές είτε ανήκουν σε ιδρύματα ή έχουν κάποιους ονομαστικούς, εκατόνομα δηλαδή μετόχους ή διευθυντές και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο απότερος πραγματικός κύριος των ε, δομών αυτών. Προσπαθήσαμε λοιπόν να εντοπίσουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δομές. Αναζητήσαμε δηλαδή τους ιδιώτες εφόσον υπάρχουν τέτοιοι και θεωρούμε αυτούς τους ιδιώτες ως απότερους πραγματικούς κυρίους. Μπορεί βεβαίως να είναι διορισμένοι κάποιοι πληρεξούσιοι οι οποίοι να εμφανίζονται και να μην εμφανίζεται ο πραγματικό κύριο. Για την ώρα αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Εξετάζοντας το που βρίσκονται τα πρόσωπα αυτά βλέπουμε ότι πάνω από τους μισούς είναι στην ε, Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό. Περίπου 8% έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σχετικά περιορισμένο ποσοστό, αλλά παρόλα αυτά είναι το τετραπλάσιο από το μερίδιο της Βόρειας Αμερικής, δηλαδή Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών αν εξετάσουμε ένα επίπεδο βαθύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουμε ότι πάνω από τους μισούς πραγματικούς κυρίους έχουν έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο και Γαλλία. Για το Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο ενδέχεται να υπάρχει κάποια διασύνδεση εκεί λόγω ρυθμίσεων ε, προξενικών θεωρήσεων για να μπορούν να διακινούνται τα πρόσωπα αυτά. Έχουμε την υποψία αυτή βασισμένη σε ονόματα, αλλά δεν γνωρίζουμε βέβαια στοιχεία διαβατηρίων κλπ. Ίσως αυτό είναι ένα ίχνος που μπορείτε να ακολουθήσετε. Ο στόχος για τον οποίο δημιουργούν τις υπερπόντιες αυτές δομές οι πραγματικοί κύριοι ή επιτρέπουν στους συμβούλους να τις δημιουργήσουν, βλέπουμε ότι εκτός από την νομοποίηση παρανόμων κερδών κλπ. που έχετε συζητήσει και εδώ στην Επιτροπή σας, πολλές από τις δομές αυτές φαίνεται βασισμένη στα έγγραφα Παναμά, καθώς και σε άλλα, χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη ή προστασία περιουσιακών στοιχείων, καθώς επίσης και για εγκληματικές δραστηριότητες. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις διαφθοράς, άρα ξεπερνά την απλή νομιμοποίηση παράνομων κερδών. Αυτό είναι το βασικό, νομίζω, συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να συγκρατήσετε από αυτήν την υπόθεση των πραγματικών κύριων. Έρχομαι τώρα στον ρόλο των ε, συμβούλων και ενδιαμέσων. Βλέπουμε εδώ βασικά τέσσερις διαφορετικές φάσεις όπου δραστηριοποιείται ο σύμβουλος ή ενδιάμεσος. Σε ορισμένε περιπτώσεις κάτι που είναι σημαντικό είναι ότι οι ρόλοι αυτοί μπορούν να αναλαμβάνονται και από τον ίδιο τον πραγματικό κύριο ή μπορούν να τον αναλάβουν επαγγελματίες οι οποίοι είναι αυτορυθμιζόμενοι. Δεν σημαίνει δηλαδή, δεν υπάρχει δηλαδή νομοθεσία η οποία επιβάλλεται σε αυτούς. Γι' αυτό το λόγο και για να καταστεί σαφές ε, ποιο είναι το ουσιώδες πραγματικά στοιχείο εδώ στον ρόλο των ενδιαμέσων, αυτά τα τονίζουμε με παχαία στοιχεία για να φαίνεται ποια είναι τα πιο ουσιώδη σημεία όλης αυτής της διαδοχικής σειράς των γεγονότων. Στις τέσσερις φάσεις λοιπόν, που είναι η συμβολή, η δημιουργία, η συντήρηση και επιβολή, βλέπετε στην φάση της συμβουλής, βλέπετε η χωρίς των συμβουλών στον πραγματικό κύριο, από τον σύμβουλο ή ενδιάμεσο, για το πώς θα στήσει την ε, υπόθεση αυτή χωρίς συμβουλών δηλαδή για επενδύσεις και τα σχετικά με επιστολές από ορκωτούς λογιστές, από δικηγόρους κλπ. Άρα είναι πράγματα τα οποία μπορούν να εκτελεστούν μόνο από περιορισμένο αριθμό ενδιαμέσων ή συμβούλων. Αυτή τη στιγμή έχει χορηγηθεί η συμβουλή η οποία μπορεί να, ζητηθεί μετα... Ε, χορηγηθεί μετά από αίτημα του πραγματικού κυρίου. Υπάρχουν για παράδειγμα τράπεζες οι οποίες έχουν δημιουργήσει ε, συστήματα τα οποία πολλούν εντός εισαγωγικών στους πελάτες τους. Είναι δηλαδή ε, μια λύση έτοιμη την οποία προσφέρουν στον ε, πραγματικό κύριο, δεν είναι σίγουρο δηλαδή ότι αυτός πρώτος ζήτησε να του γορηθήσει η σχετική συμβουλή. Στη δεύτερη φάση που είναι η δημιουργία, αυτή περιλαμβάνει την καταχώρηση της ε, δομής αυτής Υπάρχει η φάση που λέγεται domiciliation, δηλαδή της χορήγησης μιας πραγματικής διεύθυνσης στην ε, υπερπόντια κτήση, για παράδειγμα. Αυτό δεν είναι αναγκαίο για όλες τις ε, δομές, τις υπεράκτητες δομές, αλλά εκεί περιλαμβάνονται και κατόνομα διευθυντές ή επίσης μέτοχοι. Στην ουσία όλο το, το μόνο που χρειάζονται οι οντότητες αυτές είναι ένας τραπεζικός λογαριασμός. Αυτό πρέπει να θυμάστε. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί η δομή αυτή, θα πρέπει βέβαια να συντηρηθεί. Αυτό μπορεί να το αναλάβει την διαχείριση δηλαδή της ε, εταιρείας αυτής ο σύμβουλος ή μπορεί και ένας κατόνομα διευθυντής. Χρειάζεται και κάποια διοίκηση και αυτό γίνεται συνήθως από εταιρείε trust. Επίσης οι διάφορες φορολογικές εκθέσεις. Πολύ συχνά για τις δομές αυτές, αυτές δεν χρειάζεται να υποβάλουν εκθέσεις λογιστών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι θελοντικό, δηλαδή ορισμένοι από τους εμπειρογνώμονες δεν είναι αναγκαίοι. Άρα μπορεί κανείς και να το αποφύγει έρχομαι στην τέταρτη φάση που και αυτή είναι κατά κάποιο τρόπο προαιρετική. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες από πρεπόντιες ή εγχώριες δομές σχετικά με την νομιμότητα και εφόσον αυτή αμφισβητηθεί μπορεί να χρειαστούν να προσφύγουν στο δικαστήριο και στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εκπροσωπηθούν από κάποιον σύμβουλο στην πραγματικότητα συνήθως δικηγόρο. Ε, οι δικηγόροι παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. Εν τέλει, τι είδους εμπειρογνωμοσύνη χρειάζεται για να στήσετε αυτές τις επιχειρήσεις και νομική και φορολογική και λογιστική. Επομένως υπάρχουν πολύ διαφορετικοί σύμβουλοι και ενδιάμεσοι οι οποίοι διαθέτουν την ε, εμπειρογνωμοσύνη αυτή. Στη μελέτη μας εξετάσαμε τις βασικές κατηγορίες συμβούλων και ενδιαμέσων. Θεωρούμε συμβούλους ιδίως τους επιμέρους εκείνους επαγγελματίες οι οποίοι διαθέτουν τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη. Αυτοί μπορεί να ε, ε, υπόκειται σε νομοθετική ρύθμιση, μπορεί και όχι. Υπάρχουν και πολλοί εμπειρογνώμονες που δεν είναι καν μέλη αυτορυθμιζόμενου σώματος. Για παράδειγμα, οι λογιστές, οι ορκωτοί ελεγκτές, που είναι διαφορετικές οι ρυθμίσεις. Μόνο σε λίγες περιπτώσεις, σε λίγες χώρες δηλαδή. Δεν θα πω σε πολλές λεπτομέρειες εδώ, διότι ο συνάδελφός μου, Ιαν Λόξαν, θα τα πει αυτά στην ε, ε, παρουσίαση που θα ακολουθήσει την δική μου. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι οι εμπειρογνώμονες αυτοί παίζουν και τον ρόλο ενδιαμέσων. Βλέπετε εδώ ότι πολλοί ενδιάμεσοι έχουν πολυσχηδείς ε, δραστηριότητες η εμπειρογνωμοσύνη και ιδίως αυτές που χρειάζονται για να δημιουργηθούν αυτές οι υπερπόντιες δομές. Να με επιτρέψετε να έρθω τώρα στους συμβούλους. Οι πραγματικοί κύριοι λοιπόν χρειάζονται πληροφορίες για νομικά θέματα, φορολογικά, λογιστικά και επενδύσεις για να μπορέσουν να λάβουν τις ορθές αποφάσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές από, τις, πολλοί από τους συμβούλους αυτούς χορηγούν συμβουλές για πολλές και διαφορετικές πτυχές Χρειάζεται να βρουν και ενδιαμέσους, δηλαδή διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να είναι ε, προσωπικό, διοικητικό προσωπικό τραπεζών, μπορεί να είναι όμως και ανεξάρτητοι. Και διαθέτουν διαφορετικών ειδών εμπειρογνωμοσύνη, ανάλογα με τη χώρα, το νομικό πλαίσιο και ούτε καθεξής. Και είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν είναι ρυθμισμένη δραστηριότητα αυτών των ενδιαμέσων, αν θέλετε δηλαδή να στοχεύσετε σε αυτούς τα μέτρα πολιτικής. Πέραν τώρα των διαφόρων επαγγελματιών που εμπλέκονται, είναι σημαντικό να εξεταστεί και ο τόπος που έχουν την έδρα τους, διότι βλέπουμε ότι πολλοί από τους ενδιαμέσους που χορηγούν συμβούλους ιδίως, χορηγούν συμβουλές μάλλον, ιδίως σε ε, Ευρωπαίους υπηκόους έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που κάνει πολύ δύσκολη την ρύθμιση των δραστηριοτήτων τους για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η ενδιάμεση τώρα. Οι σύμβουλοι αυτοί, οι επαγγελματίε σύμβουλοι εργάζονται πολύ συχνά σε εταιρείε ενδιαμέσων, για παράδειγμα δικηγορικές εταιρείε, λογιστικές, ε, καταπιστευματικές ή τράπεζες. Και συχνά δείχνουν τα έγγραφα Παναμά για κάθε υπερπόντια οντότητα και τον πελάτη και αυτοί που συμμετείχαν στην Μοσάκ Φωνσεκά και ποιος ήταν ο ενδιάμεσος που χρησιμοποιήθηκε. Τώρα, για το πού έχουν την έδρα τους οι ενδιάμεσοι αυτοί, βλέπουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κεντρική Ασία, καθώς και Ανατολική Ασία και χώρες του Ειρηνικού. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπετε ότι περίπου 13% των ενδιαμέσων έχουν την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι περισσότεροι στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λουξεμβούργο και στην Κύπρο. Εκεί είδαμε ότι είναι κατεστημένοι και οι περισσότεροι από τους πραγματικούς κυρίους και γι' αυτό έχουν αναπτυχθεί και αυτές, αυτή η κλάδη παροχής ε, τέτοιων υπηρεσιών. Κυρίως δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες λογιστών διευκολύνουν τις ε, τη δημιουργία των ε, υπερπόντιων δομών. Αν εξετάσετε τώρα τα διάφορα δεδομένα από τα έγγραφα Παναμά, θα δείτε ότι και άλλες όπως trust companies, οι χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δραστηριοποιούνται ομοίως. Πάλι αυτά δεν έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο επαναλαμβάνεται σε ολόκληρη την παρουσίαση. Είναι δύσκολο λοιπόν να πιαστούν ορισμένοι από αυτούς ενδιαμέσους. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί οι ενδιάμεσοι. που φέρνουν ιδίως στην φάση της συμβουλής όπως εξήγησα προηγουμένως. Μονσάκ Φονσεκά, όπως είδατε, είναι, είναι υπεύθυνη περίπου για το 10%. Είτε έχουν έτοιμα συστήματα στο ράφι, δηλαδή, τα οποία πολλούν στους επενδυτές, ή τους εκπροσωπούν σε διάφορες χώρες μέλη, υπάρχει και άλλο των καταπιστευμάτων δηλαδή, άλλος ε, τομέας. Αλλά δεν καλύπτουν ορισμένες δικαιοδοσίες. Είδαμε και πριν ότι η Μοσάκ Φονσεκά εξειδικεύεται σε τρεις μόνο δικαιοδοσίες και υπάρχουν και υποστηρικτικές υπηρεσίες, κάτι το οποίο κάνουν τα τράστη δηλαδή διαχείριση, ε, παροχή ε, ανθρώπων που αναλαμβάνουν τι ευθύνε κατ' όνομα και ούτε καθεξής. Και υπάρχουν τέλο και τα χρηματοπιστικά ιδρύματα που ιδίω είναι τράπεζε αλλά και ασφαλιστικέ εταιρείε και 17% τελικώ από τους ε, μικρότερου ενδιαμέσου δεν καταφέραμε να ε, δούμε τι χαρακτήρα έχουν. Και το τελευταίο πράγμα που έχω να πω για εδώ την διαφάνεια είναι οι μεγάλες τέσσερις επιχειρήσεις, λογιστικέ λογιστικές εταιρείες δηλαδή, οι εταιρείες λογιστών, βλέπουμε από τα έγγραφα Παναμά ότι ο ρόλος εκεί ήταν σχετικά περιθωριακός, ήταν 0,15% των ενδιαμέσων. Είναι λοιπόν σχετικά περιθωριακός ο ρόλος τους. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν αυτό συμβαίνει διότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλων υπηρεσιών, άλλων εταιριών trust ή αν υπάρχουν άλλοι λόγοι και σε ποιο βαθμό Αυτές οι εταιρείες διευκολύνουν αυτή την τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Ερχόμαι τώρα στο ρόλο των τραπεζών και των ε, εταιριών Trust. Κατά τη γνώμη μας, οι τράπεζες και οι εταιρείε Trust έχουν ένα κοινό στοιχείο, ότι δηλαδή είναι ουσιώδης για ολόκληρη διαδικασία. Ο κάθε ενδιάμεσος χρειάζεται ένα τραπεζικό λογαριασμό. Και κάθε ε, υπεράκτια εταιρεία πρέπει να λάβει μορφή εταιρεία. Πώς μπορούμε να τους πιάσουμε αυτούς, διότι δεν έχουν αναγκαία την έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται. Και για τις τράπεζες ειδικότερα, εκεί υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο. Υπάρχει η νομοθεσία για την καταπολέμηση της νομοποίησης ε, παράνομων κερδών καθώς και για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης τροποκρατίας Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είναι γνωστός ο πραγματικός κύριος. Η διαδικασία, η σχετική διαδικασία διευρύνεται και βαθαίνει σιγά σιγά. Ξεκίνησε από το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος, την νομοθεσία δηλαδή για την αντιμετώπιση του, καθώς και την ε, χρηματοδότηση της το πεδίο εφαρμογή διευρύνεται για να πιάσει τώρα και την φοροδιαφυγή και αφορά αποφύγη όπως συζητούμε σήμερα. Κάποια σημαντικά στοιχεία, σύντομα λόγω χρόνου, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος εκτός από αυτό. Την νομοθεσία αυτή πρέπει να εξετάσει και το επίπεδο των ξεχωριστών δικαιοδοσιών. και τη δραστηριότητα διαφόρων τραπεζών, για παράδειγμα. Βλέπουμε εκεί ότι υπάρχει ένα σοβαρό στοιχείο συμμόρφωσης ε, με την νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Επίσης, οι πληροφορίες δεν ενημερώνονται. Άρα μπορεί να υπάρχει ένα νόμιμο μέρος, ένας, ε, ένας νόμιμος φορέας ο οποίος ανοίγει το λογαριασμό και μετά το μεταφέρει σε κάποιον παράνομο. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Εκεί πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση, να βελτιωθεί η συμμόρφωση δηλαδή με την κείμενη νομοθεσία για την αντιμετώπιση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και επίσης φορείς όπως τράπεζες μπορούν να αναθέσουν την ε, δέωσα σύνεση σε άλλους όπως η Μποσάκ Φονσεκά. Και τότε όμως πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα είναι ε, η ίδια η συμμόρφωση όπως θα το έκανε η τράπεζα. Κάτι που δεν συμβαίνει πάντοτε και πάντως όχι όπως ε, προκύπτει από τα έγγραφα Παναμά. Βλέπουμε τώρα ότι ο τραπεζικός λογαριασμός είναι ουσιώδης αλλά για να παραμείνει κλειστό το σύστημα δεν αρκεί αυτό. Χρησιμοποιούνται τώρα και εικονικά νομίσματα. Όλο και περισσότερο περνούν δε αυτά τα εικονικά νομίσματα στην πραγματική οικονομία για να αποφευθεί η ανάγκη κατοχής τραπεζικού λογαριασμού. Σε ορισμένε περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και λογαριασμοί τρίτων μερών όπως δικηγόρων, ε, λογιστών για να διατεθούν τα χρήματα στις ε, δομές offshore. Στη συζήτηση μπορούμε, αν θέλετε, να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι οι εταιρείε Trust. Mossack Fonseca ήταν δικηγορική εταιρεία, η οποία όμως είχε και άδεια λειτουργίας ως εταιρεία Trust. Μπορούσε δηλαδή να ε, δίνει μορφή εταιρεία σε διάφορες οντότητες, σε διάφορες ε, νομικές δικαιοδοσίες. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτές οι εταιρείες Trust λαμβάνουν διαφορετικά σχήματα, εξαρτάται κυρίως βέβαια από το μέγεθός τους, όσο μεγαλύτερες είναι τόσες περισσότερες υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν οι ίδιες, χωρίς να προσφεύγουν σε ανάθεση εξωτερικά και όσο μικρότερες είναι τόσο περισσότερο στρέφονται σε πελάτες με μονομένα άτομα και λιγότερο σε εταιρείες. Οι εταιρείε Trust από την άποψη της πολιτικής αυτό για το οποίο είναι σημαντικές, ε, ε, σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι έχουν την έδρα τους εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και επομένως δεν είναι δύσκολο να στοχευθούν για ευρωπαϊκές πολιτικές. Παρόλο που καλύπτονται από τις προβλέψεις της νομοθεσίας για, την, για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος και την καταπολέμηση της ε, χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Τέλος, ο ρόλος των δημοσίων αρχών υπάρχουν πραγματικά πλεονεκτήματα ε, υπέρ των διαφόρων δικαιοδοσιών για να συμμετάσχουν στα ε, διάφορα ε, συστήματα υπεράκτιων εταιριών, δηλαδή είναι και ίσπραξη φόρων, τελών για την καταχώρηση εταιριών, ανάπτυξη του τομέα των υπηρεσιών. Οι υπεράκτιες δομές δεν πληρώνουν φόρο, ό,τι είναι υποχρεωμένες να προσλάβουν κανένα. Χρησιμοποιούνται για αλλοδαπές δραστηριότητες, το οποίο σημαίνει εν τέλει ότι οι δικαιοδοσίες αυτές δεν χρειάζονται και να συλλέγουν πληροφορίες για τις υπερπόντιες δομές. Ενώ οι δικαιοδοσίες, οι εγχώριες δικαιοδοσίες, on-shore δηλαδή, έχουν το συμφέρον να συλλέγουν τέτοιες πληροφορίες. Βέβαια, είναι σχετικά απίθανο να χορηγήσει πληροφορίες αυτές mm. ο πραγματικός κύριος. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαρίστω να τις θέσετε στη διάρκεια τη συζητήσεω. Έχω μια τελευταία διαφάνεια. Συστάσεις πολιτικής. Αυτές κάπως ε, προέκυψαν και στη διάρκεια της παρουσίασης. Το πρώτο είναι το ερώτημα τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενθαρρύνει τους συμβούλους και τους ενδιαμέσους να καταπολεμήσουν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπορεί να ξεκινήσει από το ε, ε το ήπιο δίκαιο, soft law δηλαδή, μέχρι και το πλήρες δίκαιο, το οποίο προβλέπει δηλαδή κυρώσεις. Αυτά θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε στη συζήτηση με περισσότερες λεπτομέρειες. Εξετάζοντας τις διάφορες, ε, τις ενδιαμέσους και συμβούλους, Αυτές που είναι, εκεί που είναι πιο σημαντικοί οι σύμβουλοι και ενδιάμεση είναι εταιρείε trust και τράπεζες, εκεί μπορεί να ενισχύσουν την αντιμετώπιση της νομοποίησης παράνομων κερδών καθώς και ε, χρηματοδότηση τρομοκρατίας. Βέβαια, οι περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες ασκούνται μακριά από το φως. Όσο περισσότερες δραστηριότητες αυτές βγαίνουν στο φως, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η δυνατότητα να καταπολεμηθούν οι αυτέ αυτές δραστηριότητε. Ευχαριστώ κύριε Ντεγκρούν. Επανέλθουμε σε ερωτήσεις, αλλά πρώτα πρέπει να ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης από τον Dr. Ian από το LSE. Έχει εξολογηθεί ο ρόλος όσων δουλεύουν ε, και στο Λουξεμβούργο και στον Ηνωμένο Βασίλειο για τη δημιουργία και τη διαχείριση των εξωχωρευτών εταιριών, το BPI, Παναμάς και αυτή η δεύτερη μελέτη ε, που τον καθηγητή Ρόξον εστιάζει στους συμβούλους που αναλύουν και αξιολογούν τους κανόνες για την έκθεση και την ευθύνη των διαφόρων επαγγελματιών συμβούλων και διαμεσολαβητών σε κάποιες ευρωπαϊκές και άλλες ε, χώρες. Περιμένουμε να ακούσουμε τις δικές σας συστάσεις πολιτικής, ώστε και με τους κανόνες να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της ε, φοροαποφυγής, φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος χρήματος. Έχετε το λόγο. Η μελέτη είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Επιτροπής μας. Ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο, καθηγητά. Ρόξαν. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να, πρώτα απ' όλα που μας δώσει τη δυνατότητα να καταρτήσουμε αυτή και τώρα να την παρουσιάσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω το Τμήμα Πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξή του. Και πρέπει βέβαια οπωσδήποτε να ευχαριστήσω για την καταπληκτική συνεργασία και έργο τους ε, συντάκτες μας ε, από το Accounting Department του LSE και τη συγκεκριμένη της Αϊπρία Κάματ και τον προλαλήσαντα Πίτρο ε, Ντεγκρούν που μόλις ακούσατε έχω κάπως απλουστεύσει τις διαφάνειες σε σχέση με την εκδοχή που έδωσα για μετάφραση, αλλά φαντάζομαι ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε τις διαφάνειες αυτές. Θα εστιάσω στις πιο σημαντικές από τις διαφάνειες. Πώς εργαστήκαμε. Κάναμε κάποιες μελέτες περιπτώσεων. Είδαμε μια ομάδα χωρών που περιλαμβάνονται τέσσερις χώρες μέλη της Ένωσης, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Λουξεμβούργο, Κύπρος. Δύο χώρες μάλλον δύο νομιστάξεις, ε, ε, οι βρετανικέ Παρθένε νήσι και η Ελβετία που θα μπορούσαν να περιγραφούν ως ε, φορολογική παράδειση και σε έναν βαθμό συμπεριελάβαμε τις ΙΠΑ, επειδή οι ΗΠΑ έχουν κάποια ενδιαφέροντα εναλλακτικά καθεστώτα που μπορούν να μα διδάξουν πολλά. Εδώ βλέπετε ίσως το λιγότερο ενδιαφέρον κομμάτι της μελέτες ε, που Πιο πολύ είχε να κάνει δηλαδή με του κανόνε και όχι με το τι γινόταν ουσιαστικά με τα έγγραφα του Πάνω, που είναι και το πιο συναρπαστικό κομμάτι. Είδαμε λοιπόν ότι οι κανόνε ισχύουν για του επαγγελματίε, διαμεσολαβητέ, λογιστέ, ε, επαγγελματίε ε, και ελεγκτέ ή ε, διάφοροι δικηγόροι και νομικοί μπορούσαμε να βάλουμε και τους ε, συμβολογράφους ε, και τους ε, φοροτεχνικούς, φορολογικούς συμβούλους. Κάτι που δεν ορίζεται πολύ ακριβώς, επειδή υπάρχει τελείως διαφορετική κατάσταση ανά χώρα. Ποια είναι τα βασικά ζητήματα που προέκυψαν. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβουμε ποιε είναι οι υποχρεώσει των λόγω διαμεσολαβητών, τι επαγγελματικέ και τι νομικέ του υποχρεώσει έναντι των πελατών του και σε ό,τι αφορά το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Ουσιαστικά το θέμα που ε, διατρέχει τη μελέτη είναι το ερώτημα περί ανεξαρτησίας αυτών των ελεγκτών, οι οποίοι προσλαμβάνονται για να ενεργούν εξ ονόματος των μετόχων της εταιρεία, αλλά τους πληρώνει η ίδια εταιρεία. Είναι σημαντικό λοιπόν να ενεργούν ανεξάρτητα από ε, το εκτελεστικό της εταιρεία για την αξιολόγηση. Αυτού του είδους η ανεξαρτησία ε, από τους πελάτες. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλα επαγγέλματα. Ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια με την οδηγία 2014-56, κάτω Ευρωπαϊκή Ένωση, που απαγορεύει παροχή υπηρεσιών όπως ε, παροχή φοροτεχνικών συμβουλών ε, στους ε, πελάτες και σχετικές εταιρείε και φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και κάτι τελείως διαφορετικό σε σχέση με αυτό που ισχύει σε άλλα επαγγέλματα. Καταρχάς λοιπόν θέλαμε να κατανοήσουμε τι θα πει ευθύνη για άλλα επαγγέλματα και τι θα πει ανεξαρτησία. Το βασικό στοιχείο της ανεξαρτησίας ε, είναι, ε, είναι να αποφευθούν οι συγκρούσεις συμφερόντων και να διατηρηθεί οικονομική ανεξαρτησία από τρίτους. Πώς μπορούμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι εργάζονται προς όφελος των πελατών. Στην περίπτωση των νομικών επαγγελμάτων, δικηγόρων και λοιπόν, υπάρχει και μια άλλη πτυχή που εκπηγάζει από το νομικό επαγγελματικό απόρριτο ή προνομία, ανάλογα με το πώς κοιτάμε το θέμα. Η ανεξαρτησία λοιπόν είναι ανεξαρτησία ώστε να μπορούν να ενεργούν προς το συμφέρον των πελατών τους και το στοιχείο της ευθύνης σημαίνει ότι έχουν ευθύνη απέναντι στους πελάτες. Και από τα βασικά στοιχεία βέβαια είναι η εμπιστευτικότητα που είναι κοινό χαρακτηριστικό όλων των επαγγελμάτων, αν και υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό λόγω του νομικού ε, επαγγελματικού απορρίτου για τους δικηγόρους. Και το άλλο θέμα είναι ότι αυτή η διαμεσολάβηση θα πρέπει να είναι ε, ακέραιοι, αμερόληπτοι και να δρούν ε, νόμιμα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για το επάγγελμα τα αυτά, αλλά το πώς συγκεκριμένα ε, αποκρισταλώνονται μεταξύ των διαφόρων επικελματιών των διαφόρων χωρών, αλλά και μεταξύ, μέσα στην ίδια χώρα μεταξύ των επικελματιών είναι κάτι που πρέπει να αναλυθεί. Κάτι το οποίο ανακαλύψαμε και έδωσε πολλές δυνατότητες, ε, το πάντων μας δίνει τη δυνατότητα να αποχωρήσουμε σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, είναι μια εναλλακτική άποψη για τους ειδικούς επιταφορολογικά ε, δικηγόρους και δι, από τη δεκαετία του 50. Η ιδέα ότι αυτοί οι δικηγόροι μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες τους ε, να ασκήσουν και τα πολιτικά τους καθήκοντα για να μπορέσουν να προσδιορίσουν με ακρίβεια τι φορολογικέ του υποχρεώσει. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι συγκεκριμένοι δικηγόροι δεν εκπροσωπούν τους πελάτε του αστικά, αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι διαχειριστέ τη περιουσία αυτών, είτε κατεπαστευματικοί ε, διαχειριστέ και τους βοηθούν να συμμορφούνται προ τον νόμο και να προστατεύει. Στόχος είναι και η προστασία τη ακαιρότητα του νομικού συστήματο. Ένα θεματοφύλακα δηλαδή του φορολογικού συστήματος. Το ερώτημα λοιπόν που έρχεται στο μυαλό, αυτό είναι εφικτό να το πετύχουν αυτοί οι άνθρωποι. Ο σύμβουλος δεν είναι πληροφοριοδότης ή καταγγέλων, ούτε εκπροσωπεί ένα κράτος, αλλά μπορεί για παράδειγμα να μην χοργεί ε, τις υπηρεσίες που θεωρείται ότι ε, δεν είναι σύνομες. Υπάρχει και κύκλος 230 θα επανέλθω για κάποιες φορολογικές νομοδοτήσεις. Λέω ότι μπορούν να εκδοθούν μόνο ότι η συναλλαγή θα μπορούσε να επιτύχει εάν προσβληθεί. Πιο πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο θετήθηκε ο επαγγελματικό κώδικας δεοντολογίας σε σχέση με τη φορολογία. Υπάρχει ένας ε, ανεξάρτητος φορέας και ζητήθηκε να εκπονήσει από την ε, Βρετανική κυβέρνηση ένα πρότυπο σε σχέση με την παροχή συμβουλών για το φορολογικό σχεδιασμό και ζητείτε να μην προωθείτε ο φορολογικός σχεδιασμός που θα είχε αποτελέσματα ενάντια στο συμφέρον και τις προθέσεις του Κοινοβουλίου ή θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν παραθυράκια της νομοθεσίας και πάντοτε βέβαια δεν πρέπει η νομική προνομία ή τα καταστατικά επικλιματικά πρότυπα και κανόνες να παραβιάζονται. Άρα οι φορολογικοί σύμβουλοι θα πρέπει να μην προβαίνουν σε καταχρηστικής μορφής ε, φορολογικό σχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά τώρα τις καταχρήσεις, θα πρέπει να δούμε και τα άλλα στοιχεία έλεγχου. Μέσω της νομοθεσίας, δηλαδή για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος. Έχουμε την τρίτη οδηγία το 2005, την τέταρτη ε, θα αρχίσει να ισχύει από τον επόμενο μήνα και βασίζονται και οι δύο σε συστάσεις της ε, ομάδας δράσης για τη χρηματοοικονομική δράση από τον ΟΣΑ, διεθνείς δηλαδή είναι οι και όλες οι χώρες μελετήσαμε και η υποτιθέμενη φορολογική παράτηση τις έχουν υιοθετήσει, τις έχουν προσυπογράψει. Τι σημαίνει τώρα ακριβώς ξέπλυμα χρήματος. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη έννοια από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έχει τρία στοιχεία. Ευαγγελματικές δραστηριότητες, από αυτές παράγεται πλούτος και το ξέπλυμα χρήματος κατά κάποιο τρόπο είναι μια ενέργεια για την κάλυψη, κάλυψη είτε της προέλευσης είτε της ίδιας αυτού του περιουσιακού στοιχείου είτε της δραστηριότητας που κρύβεται πίσω από αυτό το κέρδος. Αυτό είναι ο ευρύς ορισμός. Ένα βασικό στοιχείο όμως είναι ακριβώς αυτή η ιδέα της εγκληματικής δραστηριότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εγκρίνει στη ε, στάση στην επιλογή ώστε να ορίζεται αυτό σοβαρό έγκλημα τουλάχιστον ε, κάθερξη ενός έτους με αυτό τιμωρείται αυτή η κλιματική δραστηριότητα τουλάχιστον. Μετά το 2012 και τις συστάσεις της ΦΑΤΦ στην τέταρτη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκάθαρα θα περιλαμβάνονται φορολογικά εγκλήματα που φτάνουν σε αυτό το όριο δηλαδή ε, σοβαρά δικήματα, predicate offenses, που είναι η βάση για αξιόπινες ενέργειες, για κλιματικές δραστηριότητες. Υπάρχει βέβαια και ένας περιορισμός. Ποια, μια επιφύλαξη, ποια είναι τα φορολογικά κλίματα, τα πιο χαρακτηριστικά που μπορεί να επηρεάζουν τέτοιου είδους συναλλαγές. Η φοροαποφυγή αφορά αποφυγή των εγχώριων φόρων κυρίως φοροποφύγει σε μια χώρα ουσιαστικά είναι το παράπτωμα το να μην πληρώνει κάποιος φόρους στη χώρα αυτή. Δεν ξεκάθαρο λοιπόν ότι αν φοροποφεύγει σε μια άλλη χώρα ή αν φοροδιαφεύγει σε μια άλλη χώρα κάποιος αυτό ε, θεωρείται και ξέπλυμα χρήματος. Βέβαια, οι οδηγίε λένε ότι η εγκληματική δραστηριότητα περιλαμβάνει εγκληματική δραστηριότητα σε άλλη χώρα. Αλλά πάντα θα πρέπει αυτό να εμπίπτει και στον ορισμό του αδικήματος, που είναι πιο περιοριστικός ορισμός σε σχέση με το ποια είναι η δραστηριότητα στο εξωτερικό που θα μπορούσε να ε, θεωρείται ως εγκληματική δραστηριότητα με βάση τις συστάσεις της ΦΑΤΦ. Η κλιματική δραστηριότητα σε μια τρίτη χώρα είναι δραστηριότητα η οποία θα πρέπει να θεωρείται κλιματική και στην τρίτη χώρα και στη χώρα που εφαρμόζει κανόνες για το ξέπλυμα, κατά του ξεπλήματος χρήματος. Αυτό το θέμα λοιπόν του φορολογικού εγκλήματος μπορεί να αποτελέσει τη βάση, ε, να είναι σημαντικό αδίκημα και θα επανέλθω στις συστάσεις. Now, the, EU e directives impose Στις οδηγίες ε, επιβάλλονται υποχρεώσεις στους ελεγκτές, ε, στους συλλογιστές, στους νομικούς, στους τεχνικούς μόνο όταν έχουν να κάνουν με διαχείριση περιουσίας, συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων ε, εντάσσονται και τα νομικά, όλα τα νομικά επαγγέλματα. Αλλά περιλαμβάνονται και αναφέρονται στο προήμιο οι φοροτεχνικοί ε, από τα νομικά επαγγελματά. Πρέπει λοιπόν να ε, εφαρμόζουν τη δέωσα επιμέλεια και, όταν, για τους πελάτες και για τους πραγματικούς δικαιούχους, να αναφέρουν τις υποψίες για εγκληματική δραστηριότητα χωρίς όμως να αποκαλύπτουν ε, τις αναφορές αυτές στον πελάτη. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που ισχύει το νομικό απόρριτο, το επαγγελματικό απόρριτο. εκτός να στηρίζει ο νομομαθής αυτός, ο νομικός αυτός την εγκληματική δραστηριότητα. Και στην τέταρτη οδηγία ε, οι φορείς αυτοί θα πρέπει να κρατούν ε, αρχεία των πραγματικών δικαιούχων, ιδίω ε, σε περίπτωση που χρειαστεί μετά να γίνει έρευνα δέωσης επιμέλειας είναι σημαντικές οι συστάσεις και απαιτήσει, αλλά θα μπορούσαν να έρχονται σε αντιπαράθεση με τη συγκεκριμένη αυτή ευθύνη αλλά και την ανεξαρτησία των επαγγελματιών. Φυσικά θα πρέπει να αναφέρονται οι υποψίες χωρίς να αποκαλύπτουν στον πελάτη. Αυτό μπορεί να έρθει σε αντίθεση, αντίφαση με την υποχρέωση του δημοσιολαβητή να ενεργεί προς όφελος του πελάτη και μπορεί να υπάρξει και σύγκρουση συμφερόντων. Βέβαια, στα επαγγέλματα αυτά ισχύουν κάποιοι κώδικες δεοντολογίας και έχουν συνταχθεί πάρα πολύ προσεκτικά για να περιλαμβάνουν και τους κανονισμούς περί ξεπλήματος χρήματος. Άρα δεν μας ανησυχεί ιδιαίτερα το θέμα αυτό. στρέφομαι σε αυτά τα επαγγέλματα που είδαμε, ελεγκτές, λογιστές, ε, τα περισσότερα ε, αυτορυθμίζονται, ε, Υπάρχουν στι περισσότερε χώρε κατευθυντήριε γραμμέ για την ε, συμπεριφορά τους, Υπάρχουν εποπτικέ αρχές για να βλέπουν να ε, και οι απαιτήσει είναι πιο λιγότερο αυστηρές στις χώρες που λέγονται καλούνται ευρωπαϊκή παράδειση. Στις περισσότερες χώρες οι λογιστές μπορούν να παρέχουν φορολογικές σύμβουλες με την επιφύλαξη των ε, ισιών των, στην σχετική, των, προβλέπει σχετική οδηγία. Υπάρχουν φορείς που προσφέρουν επαγγελματικά προσόντα. Μπορείτε να δείτε εδώ κάποια στοιχεία για κάποιες συγκεκριμένε χώρες, όπως τη Γερμανία. Μπορούν να υπάρχουν φορολογικές συμβουλές, για παράδειγμα, ή ελεγκτές, αλλά βέβαια αυτά θα αλλάξουν ε, για να προσαρμοστούν στην οδηγία τη νέα. Το Λουξεμβούργο Γνωρίζουμε ότι είναι φορικό παράδεισο, αν με επιτρέπετε να το πω. Λίγε είναι οι απαιτήσει ότι αφορά εξαρτησία και την ευθύνη και ο φορικό σχεδιασμό και συμμόρφωση είναι οι βασικέ υπηρεσίε. Υπάρχει πλήρης σχεδόν ε, στην πράξη κατάργηση του τραπεζικού απορρίτου, όμως προσπαθεί ε, να προστατεύσει αυτό το απόρριτο του Λουξεμβούργο. Είδαμε τις δράσεις κατά των καταγγελόντων ε, και στα έγγραφα LuxLeaks όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται και που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα πολλούς όπως και εμένα προσωπικά. Η Κύπρος, κέντρο επενδύσεων για χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κυρίως μπορούν να παρέχουν καταπιστωματικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σε τρίτες χώρες, οι ελεγκτές και οι λογιστές. αλλά θα πρέπει να ελέγχονται υποχρεωτικά οι, καταστα... οι εκθέσεις οικονομικής κατάστασης από ελεγκτές. Στην Ελβετία υπάρχει το λεγόμενο TESCM, Tax Efficient Supply Chain Management. Βλέπετε σε αυτό το έγγραφο τι λέει ότι σας βοηθούμε να αντιμετωπίσετε τις ανάγκες επιβολής, αποκάλυψης και με αυτή την πρακτική τεστ μπορούμε να επιτρέψουμε να πάρετε, να έχετε ωφέλη τα οποία δεν θα μπορούσατε να είχατε στην αρχή κτλ. κτλ. Στι Παρθένες νήσου, που και αυτές θεωρούνται φορολογικός παράδεισο, όπως είδαμε και στα έγγραφα του Παναμά. Μέσα σε δύο-τρει μέρε μπορεί κανεί να ιδρύσει μια εξωχωρία εταιρεία. Δεν υπάρχει νομική κατοχήρωση για τον ελεγκτή ή τον λογιστή. Υπάρχει μια ε, πράξη νομική η οποία έχει προταθεί από το 2015, αλλά δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Αυτά είναι κάποια βασικά στοιχεία και τώρα θα ήθελα να έρθω στην εφαρμογή, την επιβολή αυτών των κανόνων ε, στους επαγγελματίες. Πρώτα απ' Α, συγγνώμη. Για τους φορολογικούς συμβούλους, ε, για τους φοροτεχνικούς. Ε. Δεν ορίζεται ξεχωριστά, ως ξεχωριστό επάγγελμα στις περισσότερες χώρες. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, και σε κάποιες άλλες χώρες ορίζεται ξεχωριστά αυτό το επάγγελμα. Άλλες χώρες όμως, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν ένα εθελοντικό σώμα ε, χωρίς καταστατικές υποχρεώσεις, αλλά κώδικα διοντολογίας έχουν δικό τους. Όταν μιλάμε για εθελοντικό ε, σώμα ή για αυτούς που αυτορυθμίζονται, υπάρχει σίγουρα ένας φορέας ο οποίος ε, ρυθμίζει τη λειτουργία του επαγγέλματος, προτείνονται πρόστιμα, ε, προτείνονται μέχρι και η αναστολή της άδειας ή ε, η διαγραφή ενός μέλους. Τώρα πώς αποτελεσματική είναι αυτή η φορής, ε, ρυθμιστική φορής, δυστυχώς λίγα γνωρίζουμε. Λίγες είναι οι πληροφορίες που έχουμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας, ό,τι αφορά την παροχή φορολογικών συμβουλών. Για τους ε, λογιστές βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πρόστιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά στις Βρετανικές Παρθένες νήσου δεν υπάρχουν ε, εγχώροι ρυθμιστικοί φόροι. ό,τι αφορά του δικηγόρους βρήκαμε ότι υπάρχει σημαντική δραστηριότητα επιβολή ομοθεσίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, για άλλες χώρες δεν βρήκαμε πληροφορίες. Ε, αυτορύθμιση έχουμε στις Βρετανικές Παρθένες στο άλλο άκρο. Προβλέπονται πειθαρχικοί φορείς ε, για τους ε, δικηγόρους, δύο τον αριθμό, αλλά δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί τα μέτρα που εγκρίθηκαν πριν δύο χρόνια. Υπάρχει και κάποια ρύθμιση για, τη, για το ξέπλυμα χρήματος από την Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών που επέβαλε ποινή 400.000, 400.000 ε, δολαρίων στην Mossack ε, Fonseca το 2016. Για τους φοροτεχνικούς ε, υπάρχει ρύθμιση στο Ρωμένο Βασίλειο, αλλά είναι θελοντική. Έχουμε το 2015 54 καταγγελίες, δύο προτάσεις μορφής, μία διαγραφή και μία αναστολή δράσης. Ένα πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι τι λέει η φορολογική νομοθεσία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν κάποια καθεστώτα που μπορεί να μην είναι μοναδικά βέβαια, ισχύουν και παράνομα καθεστώτα σε άλλες ε, χώρες, αλλά στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ ανεπτυγμένο. Ντότας και Πότας είναι τα ονόματα. Disclosure of Task Avoidance Scheme, το Ντότας. Αυτή δηλαδή που προτείνουν ένα πρόγραμμα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να το αναφέρουν στις φορολογικές αρχές. Και αυτοί που το χρησιμοποιούν θα πρέπει να αναφέρουν τον αριθμό που δόθηκε στη φορολογική τους δήλωση. Υπάρχει δηλαδή εκεί ένα σημείο που αναφέρεται το κατά πόσον έχει χρησιμοποιήσει κάποιος ε, μια τέτοια, ένα τέτοιο σύστημα. Και επίσης υπάρχουν και αυτές οι ποινές, αυτά τα πρόσωπα μπορεί να φτάσουν και στο ένα εκατομμύριο αγγλικές λίρες. Ένα άλλο νέο στοιχείο είναι το λεγόμενο πότας. Αυτοί οι οποίοι δεν συμμορφούνται με τις απαιτήσει του ντότας ε, μπορεί να επισημανθούν ως πότας. και υπάρχει έντονο αποτρεπτικό αποτέλεσμα. Επίσης τα πρόστιμα ε, μπορεί να λάβει στο 100% του φόρου, φόρου που απεφεύθη ε, για επαγγελματίες οι οποίοι βοήθησαν ε, στην φοροδιαφυγή στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο πρόεδρος ενός Ιδρύματος Διαχείρισης πλούτου λέει ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι αποστασιοποιούνται από τέτοιες δραστηριότητες, αλλά η απειλή ότι θα κυνηγήσει η HMRC τέτοιους ε, συμβούλους ή οργανώσεις ε, θα έπρεπε να μας κάνει να σκεφτούμε. Συγκεκριμένο πρόεδρος της Helm Gottfried το λέει αυτό. Δηλαδή, πολλοί σκέφτονται την ευθύνη που αναλαμβάνουν και το σκέφτονται διπλά και τριπλά πριν προβούν ακόμη και στην παροχή φορολογικών συμβουλών. Άρα είναι μεγάλο το αποτρεπτικό αποτέλεσμα αυτών των καθεστώτων ιδέως για τους νομικούς. Υπάρχει επίσης μια νέα προτινόμενη νομοθεσία στο Ηνωμένο Βασίλειο, Criminal Finances Bill, ένα νομοσχέδιο λοιπόν που προβλέπει νέα δικήματα είναι πολύ πλοκοκικό αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά επειδή θα προκυρηθούν εκλογές, έχουν προκυρηθεί εκλογές, ε, τα πράγματα έχουν λίγο παγώσει και το αφήνω. Τώρα για τι Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε εδώ το καθεστώς εγκυκλίδιο 30 που σας προανέφερα, που ρυθμίζει όλου του φορεί ε, που εκπροσωπούν του ε, φορολογούμενου στο IRS, στην αρμόδια φορολογική αρχή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι, πρέπει να περάσουν τις εξετάσεις στο IRS, θα πρέπει να αποφεύγουν σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των πελατών, τυπική αρχή κατά τη σύγκρουση συμφερόντων και δεν θα πρέπει να εκπροσωπούν ιταίως υπάλληλοι του IRS ε, κάποιο πρόσωπο ε, τουλάχιστον για δύο χρόνια αφού το έχουν εγκαταλείψει την υπηρεσία τους. και υπάρχουν και κάποιες αρχές, ε, κάποια κριτήρια σε ό,τι αφορά την ευθύνη που τις βλέπετε στη διαφάνεια. Ούτε θα πρέπει να δίνουν συμβουλές εάν βασίζονται στο ότι δεν θα υπάρξει έλεγχος από το IRS. Θα πρέπει να είναι ακριβείς, άρτιες ε, οι εκθέσεις, ε, οι φορολογικές αυτές γνωμοδοτήσεις. Απλά δεν αναφέρεται συγκεκριμένα το τι πρέπει να περιλαμβάνουν. Έχει αποσυρθεί προς το παρόν λοιπόν αυτή η εγκύκλειος και είναι υπό εξέταση το θέμα. Υπάρχει και ένας ε, φορέας ο οποίος επιβάλλει τις ποινές, αλλά ας έρθω καλύτερα στα συμπεράσματα. Είδαμε λοιπόν ότι υπάρχουν παρόμοιοι κανόνε σε όλε τι χώρε, παρότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ ε, ω προ τι λεπτομέρειε. Υπάρχει ένα πρόβλημα το συντονισμό μεταξύ των κανόνων ε, όταν παρέχονται σωρευτικέ υπηρεσίε. Αυτό το οποίο χρειάζεται κατά την άποψή μας λοιπόν ένα κοινό σώμα προτύπων ε, για την παρχή φορολογικών συμβουλών για τους ε, μεσολαβητές που να συμβαδίζει με την ανάγκη προστασία του δημόσιου συμφέροντο αλλά και να σέβεται την ανεξαρτησία των επαγγελματιών. Σε ό,τι αφορά ένα πιθανό μοντέλο της εγκυκλίου 230, παρέχει κανόνες, υπάρχει ο κίνδυνος έγκρισης συμφερόντων, όταν ε, εφαρμόζονται κανόνες από τις αρχές Έχουμε τη γερμανική προσέγγιση, να υπάρχει ένα ξεχωριστό νομικά κατοχυρωμένο επάγγελμα για τους φοροτεχνικούς ε, φορολογικούς συμβούλους. Μπορεί όμως να μην περιλαμβάνει όλους τους επαγγελματίες που δίνουν συμβουλές. Έχουμε το PCRT από το Ενωμένο Βασίλειο, περιλαμβάνει τους συλλογιστές και τους δικηγόρους, αλλά ο κώδικας διοντολογίας ε, είναι ειδικά για τους ε, φοροτεχνικούς. Οι συστάσεις μας λοιπόν είναι να υπάρχει ένα ενωσιακό πλαίσιο το οποίο θα είναι ως σύσταση για την υλοποίηση των βέλτιστων πρακτικών. Θα εστιάζει δηλαδή σε επαγγελματίες που δίνουν συμβουλές ή εφαρμόζουν ενδεχομένως καταχρηστικές ε, δομές tax disclosure regimes, covered opinion rules. Θα πρέπει αυτό το πλαίσιο να ενισχύει την αξιοπιστία των κανόνων, να χρησιμοποιεί ε, τον αρμόδιο φορέα αυτό και όχι ένα αντιπροσωπευτικό σώμα. Βέβαια ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ε, καθεστώς, ένα μια νομοθετική ρύθμιση ομοιόμορφη γιατί κάθε χώρα είναι διαφορετική. Και τέλος θέλουμε να μην επιβάλλουμε υπερβολικά μεγάλες απαιτήσεις και να επιβάλλουμε την συμμόρφωση εκεί που είναι πραγματικά απαραίτητο. Έχουμε και άλλες προτάσεις να δημοσιοποιούνται τα προγράμματα φοροαποφυγής με βάση τα μοντέλα που ισχύουν σε άλλες χώρες, τα οποία μελετούμε στην Κομισιόν, να ενισχύονται οι απαιτήσει περί χρηστής διακυβέρνησης, βελτίωση διαφάνειας, η φοροαποφυγή στο εξωτερικό να θεωρείται ένα ε, φορολογικό αδίκημα που αναγνωρίζεται φορολογικό, αυτό, αυτό ως φορολογικό δίκημα και στους φορολογικούς παραδείσους. Πρέπει να γίνει κατανοητή η φύση της ανεξαρτησίας αυτών των επαγγελματιών. Είναι μεγάλη πρόκληση. Αν καταλάβουμε τις σχέσεις μεταξύ το πόσο είναι σημαντικό να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι σύμβουλοι για του πελάτε του, αλλά και ότι πρέπει να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε σημαντικέ βελτιώσει. So much, And, uh, Ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η κυρία Γκόμε. Και αμέσω τώρα έχουν το λόγο οι συνάδελφοι βουλευτέ. Πρώτα-πρώτα οι συνεισηγητέ, ο κύριο Σκόφοντ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτές τις παρουσιάσεις που είναι τόσο πλήρες και έτσι εις βάθος υπησύλθαμε στις μελέτες και να αρχίσω από την τελευταία παρουσίαση. Πολύ σημαντικές αυτές οι συστάσεις για μας. Μας είπατε ότι θέλετε να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες αυτούς. Ποια είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία που θεωρείτε ότι θα πρέπει να έχει αυτό το νομικό πλαίσιο. Πεςτε μας περισσότερο. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό αυτό το οποίο που μας είπατε σαν σύσταση, ότι θα πρέπει να αποτελεί έγκλημα το να γίνεται συνεργός σε φοροδιαφυγή ένας επαγγελματίας ή κάποια εταιρεία υπάρχει αλλά τι προβλήματα υπάρχουν ε, όσον αφορά το να προβλέπετε ένα τέτοιο έγκλημα. Τώρα όσον αφορά την πρώτη παρουσίαση, ο ρόλος των συμβούλων κλπ. Το θέμα είναι για μένα το εξή. Πώς θα αυξήσουμε την πίεση στις χώρες τις δικές μας εδώ. Πώς μπορείτε να μας προτείνετε τι να κάνουμε όσον αφορά κάποιο είδου πρότυπα, κανόνες που θα καταπολεμούν το ξέλιμα χρήματος. Εκτός μικροφώνου κυρία Γκόμες. Give the floor Πρώτα πολιτικές ομάδες οι αγορητές, πρώτα πρώτα από το ΕΛΚ. Α, όχι, όχι θα σας απαντήσουν τώρα οι προσκεκλημένοι μας και μετά κλείσουμε ομάδες έκανα λάθος, συγγνώμη. Να απαντήσω εγώ πρώτος. Όσον αφορά αυτό τον κώδικα δεοντολογίας, αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, το βασικό στοιχείο εδώ είναι η ορθή συμπεριφορά. Οι φορολογικοί σύμβουλοι σαφώς και θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές φοροδιαφυγής, αλλά για σχήματα τα οποία οδηγούν σε καταχρηστικές πρακτικές επομένως. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε ήδη και με τις υπάρχουσες οδηγίες της Ένωσης και υπάρχει εδώ η διάκριση μεταξύ αποφυγής, προσπάθειες που μπορεί να μην είναι επιτυχές και από την άλλη μεριά καταχρηστικές πρακτικές, παράνομες που μπορεί να καταπατούν ε, κάποιους δεδομένους κανόνες ε, και τελικά αντιβαίνουν στο πνεύμα της νομοθεσίας. Ήδη υπάρχουν σχετικοί ορισμοί. Σίγουρα αξίζει να διερευνηθεί αυτό για να βρούμε κάτι το οποίο αυτό θα το επεξεργαστεί καλύτερο, αλλά θέλουμε να υπάρχει ένα τέτοιο πλαίσιο για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε και να καλύψουμε το τι επικρατεί και διαφορετικά μέλη. Και το σημαντικό είναι να υπάρχει τέτοιο πλαίσιο, ούτω ώστε να έχουμε κάποια ε, ελάχιστε προποθέσει που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα κράτη-μέλη, ούτω ώστε να έχουν ό,τι του χρειάζεται σε εθνικό επίπεδο. Τώρα η άλλη ερώτηση που αφορούσε του φραγμού, τα προβλήματα όσον αφορά την παρέκταση τη ευθύνη και στις εταιρείε παροχή συμβούλου. Το βασικό εμπόδιο εδώ ότι υπάρχει δυσκολία στον ορισμό και στι ποινέ και κυρώσει που θα πρέπει να σχετίζονται με τις κυρώσεις προς τον φορολογούμενο. Στον Ιωμένο Βασίλειο έχουμε τα εξής τρία στοιχεία και προποθέσει. Θα πρέπει να υπάρχει το έγκλημα, το αδίκημα τη φορολογική από τον φορολογούμενο. Θα πρέπει να υπάρχει διευκόλυνση. Ε, Τέλο πάντων, να είναι συνεργό ο, ο επαγγελματία και να υπάρχει και κάποια εταιρεία στην οποία είναι υπάλληλο αυτό ο επαγγελματία, η οποία δεν είχε λάβει επαρκή μέτρα προστασία, αποτροπή τέλο πάντων, ή προέβλεπε κάτι και δεν το ίσκησε. Πρέπει όμως να αποδείξουν ότι είχαν μέτρα ή, ή δεν είχαν ή ότι είχαν μέτρα και είχαν λόγο να μην τα ενεργοποιήσουν. Κύριε Ντεχρούν, σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ τραπεζών και των άλλων διαμέσων, τέλος πάντων, επαγγελματιών που έχουν συμβουλές το βασικό πρόβλημα με τους περισσότερους συμβούλους, όπως είπαμε, είναι το, το, τι γίνεται όσον αφορά αυτές τις συμβουλές και βεβαίως πώς εφαρμόζεται το ισχύον δίκαιο. Τι κυρώσεις λέει, θα πρέπει να επιβληθούν. Άρα θα πρέπει να διευρυνθεί περισσότερο το θέμα. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή από τις τράπεζες και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα όσον αφορά την, τις κοινοποίησεις, την υποχρέωση των, της αναφοράς των συναλλαγών και εν προκειμένου οι υποπτικές αρχές θα πρέπει να διευκολυνθούν να ασκούν πιο δυναμικά το ρόλο τους τέλο πάντων, να επιβάλλουν αυτή την υποπτή επί των ενδιαμέσων. Τώρα κάτι άλλο είναι οι, τρά, τράπεζες πέραν των λογαριασμών που βοηθούν για κάποιο είδους εμβάσματα προς τις χώρες όπου έχει την έδρα της η εξωχώρια εταιρεία αυτή τέλος πάντων η περάκτια. Και εδώ πρέπει να υπάρχει εδώ πέρα και επιβολή, υποχρέωση, τέλο πάντων συνεργασία με τι πρωτοβουλίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριο Νίντερμαγερ, ευχαριστώ. μεστές πολύ αυτές οι εισηγήσει με πολλά τεχνικά στοιχεία. Αλλά για να σταθώ σε κάποια σημεία που είδα ότι υπάρχουν προβλήματα. Πρώτα πρώτα, ο κύριος Ντεχρούν μας είπε για τράπεζες σε σχέση με όσο είπε ο κύριος Κόφοντ. Από ό,τι κατάλαβα, θεωρείται ότι η εφαρμογή του κανόνα του να ξέρει στον πελάτη δεν αρκεί. Και επίσης, τι γίνεται τι όρια υπάρχουν, πώς επισημαίνεται ο πραγματικός, δικηγός πραγματικός κύριος, αρκεί αυτό, αρκεί το να έχουμε κάποιο κατόφλι, κάποιο όριο, να είναι δηλαδή τόσο υψηλό, ούτως ώστε να βοηθάει. Τέλος πάντων, αν μπορείτε πέστε μου, τι γίνεται με αυτούς τους λογαριασμούς υπερτρίτου. τρίτου. Πολλές φορές είναι για τον πλήρε εξούσιο, δικηγόρο, αλλά πολλές φορές αυτό διευκολύνει πληρωμές. Επίσης, μας αναφέρατε για αυτή την αδειοδότηση του να υπάρχουν εταιρείε διαχείρισης σε κάποιες χώρες. Σε ποιο βαθμό υπάρχει συμμόρφωση με τις υποχρεώσει τους, γιατί φυσικά και έχουν τεθεί κάποιες υποχρεώσεις για να μπορεί κανείς να ιδρύσει τέτοια εταιρεία. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο καθηγητή, έχω δύο ερωτήσεις για σας πρωτα Πρώτα-πρώτα, μας είπατε για την Αμερικανική νομοθεσία ότι το κριτήριο ότι η δοκιμασία είναι να το νομοθέτημα να πιάνει τόπο. Τι να πω. Τι είναι, 51-49% οι πιθανότητες του να περάσει από το Κογκρέσο και, να εφαρμοστεί, και τελικά να εφαρμοστεί. Να πείσει, να είναι πιστικό τέλο πάντων από του επαγγελματίε. Επίσης, μας ότι είναι πολύ αυστηρό το Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τα Virgin Islands εκεί όπου σχεδόν τίποτα δεν επιβάλλεται. Άρα, τελικά ποιο είναι το αποτέλεσμα όσον αφορά τους όχι και τόσο έντιμους που θέλουν να παρακάμψουν τον νόμο και να φοροδιαφύγουν. So, ευχαριστώ. Νομίζω ότι έχουμε τέτοια προσέγγιση για να καταπολεμήσουμε το, το, το, χρήματος. Πώς εκ των υστέροβε παρεμβαίνει ο νόμος. Οπότε λέμε και το κριτήριο της δέουσας επιμέλειας Τη ευξημένης επιμέλεια θα έπρεπε να ισχύει. Να, ποιο είναι το πνεύματρο όσον αφορά την κυριότητα, των το πραγματικό δικαιούχο, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Δεν υπάρχει θέμα να εγγράφεται σε ένα τέτοιο μητρό πραγματικό κύριο. Και να υπάρχει υποχρέωση δημοσίευση αυτού του μητρού. Οπότε πολλές φορές όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση έχουμε 5-6 τέτοιους κυρίους και ενδεχομένως αυτά τα κατόφληφτα τα όρια ίσως βοηθούν στον υπάρχουν παραθυράκια και έτσι να βοηθούνται ε, και άλλες εταιρείες να συσταθούν. Τώρα για την εποπτεία στις διάφορες χώρες ήδη τα έχουμε συζητήσει και ο συνάδελφος εδώ με διάφορους νομικούς. Υπάρχει διαφορετική νομοθεσία σε κάθε χώρα, οπότε σε ποιο βαθμό μπορεί κανείς να έχει λογαριασμό υπερτήρου για τέτοιες ε, δραστηριότητες. Ε, και αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα. Πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω τώρα για το τι γίνεται με την Μόσακ άκουσα τι έγινε μάλλον στον αφορά το κατά πόσο συμμορφώθηκε με τη σχετική νομοθεσία για τι εταιρείε διαχείριση για τα, για τα Virgin Islands, τον Παναμά κλπ. Ακόμη υπάρχουν τέτοια θέματα που επιλύονται ενώπιν των δικαστηρίων, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες. One minute, yes, certainly. Um... Όχι ο καθηγητής Ροξάν, καταλαβαίνω ότι σας απασχολεί το κατά πόσο είναι στέρεα τα κριτήρια στην Αμερική, αλλά πριν υπάρξει αυτό το κριτήριο, αυτός ο κανόνας, οι σύμβουλοι έδιναν το πράσινο φως όταν είχαμε πιθανότητα να πιάσουμε από το νομοθέτημα 25-30%. Άρα έχουμε προχωρήσει σε αυτό το μέτωπο. Τώρα όσον αφορά τον ρόλο των Virgin Islands, των Μαρθένων Νήσων, ε, οι κανόνες οι Βρετανικοί λένε ότι συνήθω δεν θα μπλεχτούν σε <clears throat> ύποπτες επιλήψιμε αλλαγή σε επαγγελματίες. Δεν μπορούν να νύψουν τα σχέδια του μετά. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι πολλέ φορέ έχουμε ω κριτήριο αυτό. Το να μην αγκαντεθεί ένα σύμβουλο για το ότι υπάρχει στο τέλο ένα πρόβλημα είναι κάτι επιλήψιμο. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λοιπόν. Και τώρα, εγώ να σας ρωτήσω πλευρά ε, σοσιαλδημοκρατικής ομάδας, να σας ρωτήσω το τι θα λέγατε. Εκείνους που λόγω επαγγελματικού απορρίτου αντιτίθενται εις την υποχρεωτική ενημέρωση των αρχών ο πλευράς τους. Και επίσης τι λέτε για το revolving doors, για το ότι κάποιος ε, αφού έχει υπηρετήσει στο δημόσιο μετά πάει σε ιδιωτική εταιρεία. Τι είναι με τους ενδιάμεσους αυτούς. Έχουμε θέμα και στην Πορτογαλία. Από το 2009 επιθετικές φορολογικέ πολιτικές και νομοθεσίες. Γιατί κάποιοι οι υπουργοί και οι υφυπουργοί που έχουν θεσπίσει τα σχετικά νομοθετήματα πάνε να δουλέψουν σε τράπεζες, ε, σε εταιρείε όπως η Ernst Young. Έχουμε δύο τέτοιε περιπτώσεις στη χώρα μου. Ο καθηγητή, ναι, όσον αφορά αυτό το φαινόμενο της μεταπίσης στον δικό τομέα, τι να σας πω, αυτή η εναλλαγή ε, είναι πολλέ φορέ χρήσιμη για τις φορολογικέ αρχές για να καταλάβουν ακριβώ αν πιάνει τόπο η πρακτική οι κανόνες τέλο πάντων. Και στις Ηνωμένε Πολιτείε προβλέπουν ε, κάποιο μεσοδιάστημα για να μπορείς κανείς να μεταπηδήσει. Και είναι σημαντικό αν υπάρχει κάποια υποχρέωση δημοσιοποίησης αυτό να τηρείται γιατί έτσι οι αρχές μαθαίνουν για ε, τα, τα, τα, σχήματα αυτά νωρίς, τόσο νωρίς, ούτως ώστε να βοηθάει αυτό και να τα απαγορεύουν. Και τώρα, ε, οπότε αυτό το οποίο ε, έχει, αυτό υποχρεώτη να δημοσιοποιηθεί είναι η θέσπιση αυτού του σχήματος, η δημιουργία του. Και η δημοσιοποίηση από τους ίδιους τους ε, ιδιώτες. Α, για, για, την, ε, για το απόρριτο. Ναι, ναι, αυτό έλεγα, ότι η υποχρέωση δημοσιοποίησης αφορά τα σχήματα και όχι τις ενέργειες των φυσικών προσώπων που ενέχονται. Οπότε έχουμε και... Το θέμα λοιπόν είναι η ύπαρξη αυτού του σχήματος και όχι η καθεαυτή παροχή πληροφοριών των συμβούλων προς τα φυσικά πρόσωπα, τους ιδιώτες. Και τώρα, λέει ο Πρόεδρος, πάμε στον κύριο Λουί Μισελ για την Άλτερ. Α, όχι γιατί ξέχασα για το ECR του κύριου Λούκα. Μπέρντ Λούκε. Θα μιλήσω γερμανικά. Ερώτηση προς τον Γκρούν, ο οποίος εξήγησε πολλά σχετικά με, τις οικονομικά, με τους οικονομικά ε, ενδιαφερομένους. Είπατε 60% σύμφωνα με τις έρευνές σας από τους πραγματικούς κυρίους προέρχονται από τον ανατολικό χώρο της ε, Ασίας, ενώ μόνο 8% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερώτηση. Αυτό αναφέρεται στον αριθμό προσώπων που μπορέσατε να εντοπίσετε, όχι όμως στο ποσοστό κεφαλαίου. Μπορείτε να ε, μας εξηγήσετε και σε ό,τι αφορά τις κεφαλαιακές ροές και μπορείτε να μου πείτε ποια είναι τα μεγέθη, ποιες είναι οι τάξεις μεγεθών. Μπορεί τότε να εμφανιστεί ότι οι διάφορες περιοχές του κόσμου εκπροσωπούνται πολύ εντονότερα από τον αριθμό των προσώπων. Δεύτερη ερώτηση, είπατε ότι υπάρχουν, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, διάφορα κίνητρα. Για παράδειγμα, απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων στην περίπτωση διαζυγίου ή στην περίπτωση νομοποίηση παρανόμων κερδών ή τρομοκρατικών ε, δράσεων. Εάν αυτές οι τόσο διαφορετικές προσπάθειες μπορούν να εξυπηρετηθούν από τις ίδιες νομικές δομές, δηλαδή τελείως διαφορετική υπόθεση αν θέλω να αποκρύψω περιουσιακά μου στοιχεία στην περίπτωση διαζυγίου και τελείως διαφορετική περίπτωση η ε, προσπάθεια χρηματοδότησης τρομοκρατικών ε, πράξεων. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, μπορεί κανείς από τη νομική δομή ε, μιας επιχειρήσεως να συναγάγει συμπεράσματα σχετικά με το ποιο σκοπό εξυπηρετούσε η ε, προσπάθεια εξόχωρης απόκρυψης. Μπορούμε να εξαγάγουμε συμπεράσματα δηλαδή από τον τρόπο που είναι δοδημένη μια συγκεκριμένη επιχείρηση ή όμιλος επιχειρήσεων. Ο κύριος Ντεγκρούν, ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Πρόκειται για ένα από τα βασικά θέματα που αντιμετωπίσαμε στην αναλυσή μας, ότι έχουμε πληροφορίες μονάχα για τον αριθμό των ε, διαφόρων οντοτήτων και όχι για το τι ακριβώς κάνουν. Υπάρχουν πολλά έγγραφα που έλαβε η αρμόδια αρχή, αλλά τα δημοσίευσε είτε μόνο για την οντότητα, για τους συνδιαμέσους που, είναι, που εμπλέκονται τους ε, ε, ε, συμβούλους και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή τόσο πολλά για τη δραστηριότητα εντός των ίδιων των φορέων. Δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να αρκεστούμε στον αριθμό των προσώπων. Βλέπουμε τον αριθμό των ε, φορέων αυτών να μειώνεται, δεν σημαίνει όμως ότι μειώνονται οι δραστηριότητες. Τώρα, κίνητρα και δραστηριότητες. Σύμφωνα με τις ε, αναφορές από του ICIJ και από τη διαρροή των ε, εγγράφων του Παναμά, νομίζω ότι είναι ενδιαφέρουσα η ιδέα. Ίσως έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε κάποιες τεχνολογίες ε, ανάλυσης δεδομένων να δούμε Δύο για περίπλοκες δομές που όπως είπατε και εσείς μπορεί να χρησιμοποιηθούν περισσότερο για την απόκριψη ε, περιουσιακών στοιχείων ή για το ξέβλημα χρήματος. Φαίνεται πως τα έγγραφα Παναμά αποκαλύπτουν μέρος μόνο της δομής. Δεν έχουμε δηλαδή αναγκαστικά όλες τις προφορίες. Ίσως μπορούμε να έχουμε κάποιες γενικές κάποια γενική ιδέα, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο να διακρίνουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται. Αλλά θα έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Okay. There was a change here. Uh, welcome to everybody. Carlos ορίσατε. Χθες ήταν η γιορτή των εργαζομένων, πρωτομαγιά. Άρα θα πρέπει να σεβαστούμε το ώρα των τερμηνέων και άρα θα πρέπει να σας ζητήσω όλοι να είστε όσο γίνεται πιο σύντομοι. Ο επόμενος ομιλητής τώρα είναι ο Λουί Μισελ από τους Φιλελευθέρους. Δεν σας υπόσχομαι θα είμαι όσο σύνος θέλετε. Γιατί άκουσα όλες αυτές τις μακρές επεξηγήσεις, αλλά πρέπει να σας ρωτήσω το εξής. Τι λέτε στην υποχρέωση των τραπεζών προς τους νομικούς και συνετικές αρχές να υπάρχει ένα δημόσιο μητρό αυτών οι οποίοι ελέγχουν τις επιχειρήσεις και άλλα νομικά πρόσωπα, δηλαδή πέραν των ε, μετόχων αυτό το μητρό θα είναι διαφορετικό από το μητρό των μετόχων και έτσι θα φαινόταν ποιοι είναι οι πραγματικοί κύριοι μια επιχείρηση. και αυτό θα έχει δημόσιο χαρακτήρα και μπορούσε όποιο θέλει να το συμβουλευτεί. Δεύτερον, η οδηγία κατά του πλησίματος λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο μητρό για ιδρύματα και εταιρείε. Τα κράτη-μέλη ε, πρέπει να το κάνω αυτό με το 2016 τον Ιούνιο, έλεγε, για να ε, νομοθετήσουν στα πλαίσια του εθνικού δικαίου. Για πέστε μας, έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία της κύρωσης, γιατί ε, από ό,τι γνωρίζουμε οι διατάξεις που διέπουν τα διαφορονομικά πρόσωπα, όπως ξέρετε, ποικίλουν πάρα πολύ από μια χώρα στην άλλη. Και τώρα και δύο πολιτικές σκέψεις μου, αγαπητοί συνάδελφοι. Θεωρώ ότι η Επιτροπή μας Σήμερα χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση συνοπτική μεν, αλλά να γίνει για το τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε όσον αφορά το θέμα των εγγράφων του Παναμά. Οπότε ή θα ολοκληρώσουμε αυτή την επιτροπή με κάτι το φιλόδοξο, με κάποια είδους βάσιμες συστάσεις, ακριβώς όπως είπε ε, ο δεύτερος εκ των ομιλητών μας, αυτό που είπε για αυτό το ε, μάξιμου και συγκεκριμένο κατόφλι και όριο που θα δεσμεύει τα κράτη-μέλη. Οπότε εμεί θα πρέπει να πιέσουμε με τέτοιου είδου όραμα τα κράτη-μέλη και με συστάσεις. Και γιατί θα πρέπει ο κόσμο να ξέρει ποιο θέλει τι εδώ στι Βρυξέλλε για αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Άρα πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή. Ή το ένα ή το άλλο. Και το άλλο είναι να συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοιου είδους ε, προτάσεις για καλύτερη συνεργασία, καλύτερες καταγγελίες, αλλά όλα αυτά να είναι μόνο λόγια. Άρα εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε και θα πρέπει να γίνει πολιτική συζήτηση για να αποφασίσουμε ποιο από τις δύο ατραπούς θα ακολουθήσουμε. Uh, two minutes left for the όμως σας έχουν μείνει μόνο δύο λεπτά. Για την ποια Για την απάντηση, Α, το, η δεύτερη ερώτηση αφορούσε την εφαρμογή της οδηγίας, της τέταρτης οδηγίας για το ξέπλυμα. Έχουν προθεσμία τα κρατημέλη μέχρι τον επόμενο μήνα έχουν υποθέτω προχωρήσει τα μελη διάφορα Έχουν έχουν θεσπίσει σχετική νομοθεσία εφαρμοστική της οδηγίας και βέβαια τον έχουμε αυτά τα μητρώα των ε, πραγματικών κυρίων αυτό θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να καταλάβουν τι υποχρεώσεις έχουν να εξασφαλιστεί ότι δεν θα διευκολύνουν τέτοιες δραστηριότητες. Τώρα όσον αφορά αυτό το μητρό, έχουμε κάποιες εταιρείες νομικά πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αποτελεσματική νομοθεσία θα πρέπει τα μητρώα να καλύπτουν και αυτές τις, αυτά τα νομικά πρόσωπα και τα πρόσωπα που εκεί εμπλέκονται και ως μέλη Συμβουλίου και ως μέτοχοι πέραν αυτών που πραγματικά ασχολούνται με την καθημερινή εταιρική δράση. Και αυτό να ληφθεί υπόψη όταν αποφασιστεί το τι θα γίνει με το σχετικό μητρό. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Από την ε, Γκουε, είναι από την ίδια πολιτική ομάδα με εμένα, οπότε του παραχωρώ τον χρόνο μου, του κύριου Μακάρθη. Α, ως συνήθως, η Γερμανία έτσι γέρονται σε εμά του Ευχαριστούμε τέλο πάντων και την ερευνητική υπηρεσία. Έχω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την μελέτη για συμβούλους και ενδιάμεσους. Πρώτα πρώτα, η γλώσσα που πολλές φορές σημαίνει ότι πολλές φορές αυτή η ενδιάμεση και η σχετική νομική βοηθούν σε τέτοιου είδους επιλήψιμα σχήματα. Η συνεργή λοιπόν σε αυτό το αδίκημα ε, καλύπτονται από την νομοθεσία στη δική μας, στην Ιρλανδία. Και προβλέπεται υποχρεωτική δημοσιοποίηση κάποιων πληροφοριών. Ίσως και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις για την πολιτική μας, για την ανεξαρτησία, την ευθύνη, νομίζω ότι πήραμε το μάθημά μας με αυτήν την έρευνα που κάνουμε όσον αφορά το τι γίνεται με τον κώδικα διοντολογίας για αυτές τις εξωχωρές δραστηριότητε. Μήπως ο κύριος καθηγητής έχει κάποια παραδείγματα από θετική εμπειρία από κάποιες καλές πρακτικές και πρωτογενές δικαιωτρά όσον αφορά τις διαβουλεύσεις μας και τις κυρώσεις τις κυρώσεις εις βάρος των επαγγελματιών όταν δεν τηρούν την υποχρέωση πληροφόρηση και δημοσιοποίηση. Ακριβώς δύο λεπτά έκανα, Πρόεδρε. Ναι, ναι, ναι, το είδα, όντως, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας, λέει ο κ. Δεχόρων. Έχουμε έναν ευρύτατο ορισμό του τι θα πει ενδιάμεσος, όχι μόνο ο σύμβουλος επομένω, αλλά και αυτός ο οποίος συμβάλλει στην ίδρυση μιας εταιρείας και στην ε, διατήρηση, τη λειτουργία της. Άρα να πούμε συνεργώς ίσως θα το στένευε. Αν θέλετε στενορισμό, ναι, αυτό που ισχύει τώρα. Όσον αφορά το θέμα ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ευθύνη. συνεργάστηκα και με τον Ιαν για το δικό του κείμενο. Οπότε κάθε επιτροπή είναι κοινέ οι προτάσεις, οι στάσεις μας. Για τα περισσότερα τα λέμε στην εκθέση του Ιαν. Άρα δεν είναι θέμα του ότι έχουμε μόνο σόφτλο, δευτερογενές ε, και μη υποχρεωτικό δίκαιο. Ρόξαν. Θέλουμε να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερους. Ακόμα για αυτούς που δεν θεωρείται ότι συμβάλλουν στο ξέπλυμα. Γι' αυτό και θέλουμε ευρύ ορισμό. Τώρα όσον αφορά την νομοθεσία, μεταξύ άλλων λέμε ότι τα, τα σώματα και οι φορείς εκπροσώπησης θα πρέπει να καλύπτονται από την νομοθεσία. Και επίσης με τις συστάσεις μας θέλουμε να καλύψουμε κάτι το οποίο μόλις τώρα ανακοινώθηκε στη ΣΥΠΑ. Ένα υποπτικό σώμα για, τα, για αυτούς τους φορείς αυτορύθμισης για το ξέπλυμα. Και να υπάρχει έλεγχος ε, ισοτήμων στον κώδικα διοντολογίας που να καλύπτει πέραν της διοντολογίας και την εφαρμογή του νόμου. Οπότε όσον αφορά την άρεστη πρακτική Έχουμε διαπιστώσει σε όσες χώρες έχουν υποχρέωση ενημέρωσης και πληροφόρησης και έχουν θεσπίσει και κυρώσεις ότι υπάρχουν επιπτώσεις όσον αφορά τη συμπεριφορά των επαγγελματιών συμβούλων. Τι γίνεται όμως με τις ξεχωριστές δραστηριότητες, όπως είπαμε. Το θέμα είναι τι ορισμό δίνει το ιστορικό δίκαιο στο φορολογικό αδίκημα. δεν έχει δίκιο παραδοσιακά λέει ότι, ότι το, το φορολογικό δίκαιο είναι εθνική αρμοδιότητα. Όμως έχουμε τις κοινοτικέ οδηγίες και άλλα στοιχεία τα οποία λένε και αυξάνονται και αυτό το προωθεί και για την αμοιβαία αρρωγή. Άρα αυτά τα διεθνή στοιχεία πρέπει να δούμε πώς θα τα ενσωματώσουμε ε, στο τι θα θεσπίσουν σαν κώδικα αντιολογίας για τους επαγγελματίες. Πασκάλ Τυρό. Πράσινο. Τρεις ερωτήσεις. Να μου πείτε τη γνώμη σας. Πρώτα πρώτα, τι γίνεται όσον αφορά το καθεστώς που διέπει τους ενδιάμεσους. Εάν τους θεωρήσουμε ως συναυτουργούς των αδικημάτων, να μην έχουμε κυρώσεις μόνο για τους πελάτες. Να, μια ιδέα για το τι να κάνουμε συναυτουργεί άπαξ και συντρέχει περίπτωση απάτης. Επίσης αυτό το οποίο είπατε όσον αφορά αυτές τις επιστολές που οδηγούν σε απαλλαγή κάποιων εμπλεκομένων γιατί καλύπτονται από αυτές τις επιστολές. Αυτού του είδους οι επιστολές επιβεβαίωσης να απαγορευτούν. Τρίτο υπάρχει απουσία ενημέρωσης για τους μονίμως διαμένοντες κάπου. Δεν παρέχουν φορολογικές ε, αρχές πληροφορίες σε κάποιον που πάει σε μια χώρα για να φτιάξει ένα τέτοιο σχήμα. Μήπως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε αύξηση των επιλήψιμων ε, συμπεριφορών και σχημάτων. Μήπως έχετε κάποια πρόταση για το πώς θα επιληθεί αυτό το πρόβλημα. Well, Απάντηση. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς των ε, ενδιαμέσων ως συναυτουργών, εξαρτάται από τι ακριβώς πράττουν. Σε ορισμένε περιπτώσεις θα είναι με τις νομοθετικές νοθήσεις που ανέφερα προηγουμένως για την ευθύνη των εταιριών. Σε ορισμένες περιπτώσεις η ευθύνη διευκόλυνσης θα εξαρτάται από την ε, ε, πρόθεση και την δράση του ενδιαμέσου. Εξαρτάται εάν οι συμβουλές που δόθηκαν είναι γενικές και αν η εφαρμογή τους αναλήφθηκε από άλλους που δεν ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι, θα είναι πιο δύσκολο να ε, χαρακτηριστεί με τον τρόπο με τον αρκετόν β' τρόπο. Αυτό είναι και ένα από τα ζητήματα που προκύπτουν από την χρήση δικτύων ενδιαμέσων. Σε ό,τι αφορά τις επιστολές προθέσεων στις οποίες αναφερθήκατε, δεν δίνονται τέτοιες μόνο για ζητήματα ε, φορολογικά. Αποτελούν ένα ε, πρακτικό νομικό εργαλείο. Υπάρχουν πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτές και ίσως ένα θέμα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τα νομικά επαγγέλματα δεν είμαι βέβαιο ότι μια αυστηρή απόφαση σχετικά με τα φορολογικά θα είναι και παραγωγική, διότι υπάρχουν πολλές φορολογικέ υποθέσει που δεν ενέχουν το στοιχείο της καταχρήσεω. και όπου τα μέρη έχουν κάποια αίσθηση της ευθύνη για τις νομικές συμβουλές που παρέχουν. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό προσώπων που έχουν διπλή ηθαγένεια Mm. Εάν αυτός ο αριθμός αυξάνει ή όχι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά νομίζω τα τελευταία χρόνια υπάρχουν περισσότερες χώρες που προσφέρουν τέτοιου είδους προγράμματα. Είναι μια παρατήρηση αυτή που κάνω οποία θα πρέπει να ελεγχθεί. Στα έγγραφα Παναμά βλέπουμε μόνο ότι υπάρχουν ορισμένες χωρισμένοι που υπερεκπροσωπούνται σε ό,τι αφορά τον αριθμό υπηκόων τους. Υπάρχουν και ορισμένα ονόματα που δεν φαίνεται να είναι ηθαγενή κάποιας χώρας και είναι προφανές ότι έχουν εγκατασταθεί εκεί από κάπου αλλού. Πρόεδρος, τεμάζει. Οι ομάδες EFDD και ENF δεν έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λάβουν το λόγο για την ώρα. Ο τελευταίος λοιπόν ομιλητής είναι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και νομίζω ότι είναι ο κ. Ρωσάτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από τα όσα μας είπατε αντιλαμβάνομαι ότι αυτοί οι ενδιάμεσοι, οι διευκολυντές υπάγονται σε ένα διτό σύστημα εξωτερικής ρύθμισης και ενδορύθμισης, δηλαδή μέσα στις οργανώσεις που οποίες ανήκουν. Και αυτό εξαρτάται από τη χώρα. Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι το σύστημα δεν είναι πολύ αποτελεσματικό όσον αφορά την πρόληψη, να προλαμβάνεται δηλαδή οι επαγγελματίες αυτοί να συμβάλλουν σε κάποιες επιζήμιες για το δημόσιο φορολογικές πρακτικές. Μπορεί κανείς να κρίνει με πολύ αυστηρό τρόπο το συνδυασμό αυτό. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας. Δυστυχώς ήρθαμε κάποια καθυστέρηση και δεν είχα την ευκαιρία να σας ακούσω από την αρχή. Αλλά ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την επιβολή πολύ αυστηρότερων νομικών υποχρεώσεων σε νομικούς συμβούλους και φορολογικούς συμβούλους για να τους απαγορευτεί στην ουσία να εμπλέκονται σε κάθε είδους φορολογικό σχεδιασμό και να αναφέρονται τέτοιες υποθέσεις στις φορολογικές αρχές εφόσον προκύπτουν. Είναι κάτι τέτοιο δυνατό να επιβληθεί στην πράξη και σε ποιο βαθμό θα μπορέσουμε έτσι να συμφιλιώσουμε την ανάγκη να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του πελάτη με την επιταγή συμμόρφωσης της νομικές νομοθετικές διατάξεις δηλαδή. Βεβαίω, σε κάθε προσπάθεια των πέλατων να μειώσουν τη φορολογική του ευθύνη είτε νόμιμα είτε παράνομα. ενδιαφέρουσα ερώτηση και μια πραγματική πρόκληση. Αναφέρεστε στο βαθμό εμπλοκή στον φορολογικό σχεδιασμό. Και τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε φορολογικό σχεδιασμό στο πλαίσιο αυτό. Σαφώς οι επαγγελματίε αυτοί δεν θα πρέπει να διευκολύνουν την ε, φοροδιαφυγή. Αυτό θα έπρεπε να είναι αυτονόητο. πολλές από τις ε, υπερπόντες αυτές τις δομές εμπλέκονται σε φόρο διαφυγή. Υπάρχουν και ενδείξεις ότι εμπλέκονται και σε φόρο αποφυγή. Υπάρχει μια άλλη ανησυχία σχετικά με τον καταχρηστικό φορολογικό σχεδιασμό σε μια προσπάθεια καταστατήγησης των φορολογικών νόμων Πολύ συχνά όταν κάποιοι υπερασπίζονται τις δραστηριότητες αυτές λένε «Μα κοιτάξτε είναι απόλυτα νόμιμο». Εμένα αυτό δεν μου φαίνεται ορθό. Διότι είναι ατελώς νόμιμες και όχι εντελώς νόμιμες. Μπορεί να είναι ή όχι αποτελεσματικές οι δράσεις αυτές. Βασίζονται στον ισχυρισμό ότι η ερμηνεία του νόμου, στην οποία στηρίζονται, είναι ισχυρά, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί βέβαια όταν θα έρθει η ώρα, αλλά βασίζονται σε έναν ισχυρισμό νομιμότητας και μου φαίνεται δύσκολο να δει κανείς από την αρχή που μπορεί να βάλει το όριο. Γι' αυτό εμείς προτιμήσαμε να προτείνουμε να διατυπωθεί ένα κώδικα διοντολογία που θα λέει στου επαγγελματίε, κοιτάξτε πρέπει να τα σκεφτείτε τα πράγματα αυτά και έχετε υποχρέωση να μην υπερβείτε το όριο, αλλά και ο ίδιο ο επαγγελματία να εξετάσει να βρει πού βρίσκεται το όριο. Και αλλιώ να ζητήσει συμβουλή από άλλου επαγγελματίε σχετικά με το πού βρίσκεται το όριο. Είναι δύσκολο να καταλήξει κανείς σε κάτι το οποίο θα είναι δυνατόν να επιβληθεί σε κάθε είδους φορολογικό σχεδιασμό. Εάν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπησέρχονται λάθρα κάποια στοιχεία φοροαποφυγής σε τέτοιες δομές, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έθιξε στην παρουσίασή του και ο Πέτερ και Αυτά που προκύπτουν από τα έγγραφα Παναμά δείχνουν πόσο σημαντικές είναι, είναι οι προφορίες για αυτά. Άρα σωστά δέτε την ερώτηση, εάν όντως είναι δυνατόν να επιβληθούν τέτοιες υποχρεώσεις και είναι πολύ δύσκολο να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση. Πρόεδρος Ντεμάζη, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο ερευνητές τον κύριο Ρόξαν του LSE και τον κύριο Ντεγκρούν και θα ήθελα την διαβεβαίωσή σας ότι εάν κάποια από τις πολιτικές, πολιτικές ομάδες έχουν, έχει κάποια συγκεκριμένη ερώτηση να μπορέσουν να την υποβάλουν γραπτός. Για παράδειγμα, ο ρόλος των δικηγόρων και πώς μπορεί να ρυθμιστεί. Να υπάρξει κάποιος τρόπος λοιπόν να επανέλθουν. Αναμένουν ε, τώρα η δεύτερη ομάδα των ερευνητών μας. Ας ε, περάσουμε αμέσως στο δεύτερο πάνελ, διότι έχουμε και μια καθυστέρηση 10 λεπτών, αλλά θα την ε, καλύψουμε. Θα ασχοληθούμε τώρα με μια μελέτη για την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου των πρακτικών εξωχώριων δομών για τις υπεράκτητες πρακτικές σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη. Έχουμε πρώτα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γκρόνιγκεν, τον κύριο Μπρόρινγκ, ο οποίος θα αναφερθεί ε, στο τι συμβαίνει στο βασίλειο των κάτω χωρών. Έχουμε μετά τον κύριο Πίτερ Κλέγκ από το Δυτικό Πανεπιστήμιο ε, στο Μπρίστολ της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και τον κύριο Μετρό Ντελαμότ του Πανεπιστημίου Κρετέι του Παρισιού, ο οποίος θα εξηγήσει τα των γαλλικών υπερπόντιων εδαφών. Θα σας παρακαλέσω να περιοριστείτε μεταξύ 12 και 15 λεπτών, θα μας βοηθήσετε πολύ έτσι. Δεν θα προχωρήσω σε Εισαγωγικέ παρατηρήσεις για να ε, εξοικονομήσουμε κάποιο χρόνο, να παρακαλέσω πρώτα τον κύριο Μπρόρινγκ να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το βασίλειο της Ολλανδίας έχει ένα ομοσπονδιακό χαρακτήρα και το νομικό του πλαίσιο είναι αρκετά περίπλοκο. 5% μόνο του Ολλανδικού πληθυσμού το γνωρίζει καν αυτό το πλαίσιο. Έτσι θα χρειαστεί μια πολυσχηδής ανατένιση που βλέπετε στην επόμενη διαφάνειά μου. Και κάθε επίπεδο αντικατοπτρίζει και ένα κεφάλαιο της εκθεσής μας. Το βασίλειο των κάτω χωρών είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται πλήρως μόνο στην γεωγραφική ευρωπαϊκή επικράτεια του βασιλείου. Το βασίλειο της, των κάτω χωρών αποτελείται από τέσσερις Αρούμπα, Κουρασάο και Άγιος Μαρτίνος και βεβαίως και την χώρα των κάτω χωρών. Η συνθήκη λειτουργίας της Ένωσης αναφέρει και τις Ολλανδικές Αντίλες που αποτελούσαν έδαφος του βασιλείου μαζί με ε, Μπονέα, Στάσια και Σάβα, αλλά από το 2010 οι Ολλανδικές Αντίλες δεν υπάρχουν πλέον. Οι τρεις καραϊβικές χώρες έχουν περίπου 150.000 κατοίκους από το 2010 όταν έγινε μια αναδιάφρωση μέσα στο βασίλειο των κάτω χωρών. Οι χώρες Μπονέα, Στάσια και Σάμπα αποτελούν πλέον μέρος της επικράτειας των κάτω χωρών, η οποία έχει ένα ευρωπαϊκό μέρος και ένα καραϊβικό μέρος, της, την Ολλανδική Καραϊβική. Από την αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλα τα νησιά της Καραϊβικής, οι Καραϊβικές χώρες, τμήματα δηλαδή του ε, Βασιλείου της Ολλανδίας έχουν χαρακτήρα OCT. Επομένως, το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται μόνο στην επικράτεια της, ε, ε, των κάτω χωρών. Το ευρωπαϊκό δίκαιο εφαρμόζεται και στις καραϊβικές χώρες, χωρίς από τις λεπτομέρειες εδώ. Αναφέρομαι στο παράδειγμα 4 τη συνθήκη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεσή μας αναφερόμαστε σε νομολογίες της αποφάσεις Antillian Rice Mills και Eman and Sevinger. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την μείωση οικονομικής βοήθειας για υπερπόντια εδάφη και χώρες. Οι νομικές εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την εποπτεία, καθώς επίσης και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Καταπολέμησης των Απατών, είναι πολύ σημαντικά. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε το προήμιο της Overseas Association Decision, OAD, που επιβάλλουν διεθνείς διατάξεις στις ε, οικονομικές υπηρεσίες. Εκεί τονίζεται ιδιαίτερο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Υπηρεσίας Καταπολεμής Απατών. το βασίλειο των κάτω χωρών αποτελείται από τέσσερις ισότιμες χώρες, επισήμως. Στην πράξη όμως κατησχύει η επικράτεια στην Ευρώπη των ε, κάτω χωρών που έχει βέβαια και τους μεγαλύτερους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι το δίκαιο των τριών χωρών της Καραϊβικής εμπνέεται σημαντικά από την ομοθεσία των ευρωπαϊκών κάτω χωρών. είναι δηλαδή ε, νομικά μοσχεύματα. Η το μεγαλύτερο μέρος της νομοθεσίας των ε, καραϊβικών χωρών της, ε, του βασιλείου των κάτω χωρών είναι πρώην Ολλανδική νομοθεσία, η οποία επειδή βασίζεται στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και ιδίως ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή, την φορολογική διαφάνεια και το ξέπλυμα μαύρου χρήματο, μπορεί να πει κανεί ότι η νομοθεσία αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Παρόλο που ε, πρόκειται για μια προηγούμενη εκδοχή του δικαίου αυτού. Η νομική κατάσταση των ε, τριών αυτών υπερπονδίων εδαφών της Ολλανδίας είναι πολύ διαφορετική, διότι καλύπτονται από τον νομοθέτη που έχει έδρα του τη Αλλά θα επανέλθω σε αυτό αργότερα η σωστή κατανόηση του θεσμικού πλαισίου του Βασιλείου της Ολλανδίας προϋποθέτει και γνώση της ευαισθησίας της σχέσης μεταξύ των δύο αυτών τμήματων που έχουν ανάμεσά τους τον Ατλαντικό. Βεβαίως έχουν μείνει ίχνη για να μην πω ε, ουλές από τη διαδικασία αυτή. Η ευαισθησία έχει βέβαια σχέση και με τις πολιτιστικές διαφορές αλλά και την έλλειψη ισορροπία στην εξουσία αρμοδιότητας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τμήματο και των Καραϊβικών Τμήματων του Βασιλείου τη Ολλανδίας. Η Ολλανδική κυβέρνηση της Χάγης είναι πολύ διστακτική σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να παρέμβει στις πολιτικές των καραϊβικών χωρών της Ολλανδίας. Για παράδειγμα στις παραβιάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας στις παραβιάσεις ε, θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που δεν αιτιολογούν παρόλα αυτά παρέμβαση στις πολιτικές μιας χώρας της Καραϊβικής, Ολλανδικής Καραϊβικής, ενώ πάντα. Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις παρεμβαίνει η Ολλανδική κυβέρνηση. οφείλει να αναγνωριστεί ότι οι καραϊβικές χώρες του Βασιλείου της Ολλανδίας είναι κοινωνίες μικράς κλίμακος και ως τέτοιες είναι δύσκολο εκεί να εκριζωθεί ο νεποτισμός και ε, μια πόλωση. Οι λαοί των χωρών αυτών της Καραϊβικής τα γνωρίζουν αυτά παρόλο που παραπονούνται για την κατήσχηση ε, των ε, δικαστών που προέρχονται από το υπηρετικό τμήμα της Ολλανδίας δέχονται τις αποφάσεις τους για την διατήρηση του κράτους δικαίου και υπέρ μιας σταθερότητας που είναι σημαντική για την οικονομία και ιδίως βέβαια για τον τομέα του τουρισμού. Ο χάρτης, ο χάρτης του Βασιλείου στο άρθρο 3 του διαλαμβάνει τις εξουσίες του Βασιλείου που περιορίζεται στην άμυνα εξωτερικά και ζητήματα ηθαγένειας. Άλλες εξουσίες του Βασιλείου είναι η δυνατότητα να ακυρώσει μια νομική διάταξη μιας καραϊβικής χώρας, καθώς επίσης και να παρέμβει εάν μια καραϊβική χώρα, της Ολλανδίας πάντα, δεν, εκπροσω... δεν ε, ε, ανταποκρίνεται στις υποχρώσεις της. Υπάρχει και το άρθρο 43, επιτρέπει να εξετάζονται και κανόνες χρηστής διακυβέρνησης. Όσον αφορά φοροδιαφυγή, φορολογική διαφάνεια και ξέπλυσμα μαύρου χρήματος, η νομοθεσία των τριών καραϊβικών χωρών επηρεάζεται σημαντικά από την νομοθεσία της, της Ευρωπαϊκής Ολλανδίας. Επομένως, κανονικά θα πρέπει να αρκεί η νομοθεσία αυτή για την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων που απορρέουν από τις δραστηριότητε αυτές. Δεν είναι βέβαια και μυστικό από την άλλη μεριά ότι στις χώρες αυτές της Καραϊβικής η εφαρμογή και επιβολή της νομοθεσίας είναι κάπως ασθενής λόγω σπάνιδος πόρων αλλά και ανθρώπινου δυναμικού και είναι ένα γενικό συμπέρασμα όταν έχουμε, ε, ότι έχουμε την εντύπωση ότι θέματα φορολογικής διαφάνειας και ε, ξέπλυματος αντιμετώπιση, δηλαδή ξέπλυματος μαύρου χρήματος κλπ. δεν έχουν πολύ ψηλή προτεραιότητα. η Ευρωπαϊκή Ολλανδία συνεργάζεται εντός του Βασιλείου και με τις ε, χώρες της Καραϊβικής. Και αυτή η συνεργασία απηχείται, για παράδειγμα, με την οικονομική εποπτεία στο Κουρασάο και τον Άγιο Μαρτίνο και με την οικονομική εποπτεία με Συμβούλιο Οικονομικής Εποπτείας. Δεύτερο, και οι τρεις καραϊβικές χώρες είναι εξοικειωμένες με την κεντρική τραπεζική εποπτεία για θέματα στοιχηματισμού, φοροαποφυγής, φορολογικής διαφάνειας και ούτε καθεξής. Και η κεντρική τραπέζα της Αρούμπα και του Κουρασάου και του Αγίου Μαρτίνου. Και οι δύο καραϊβικές τράπεζες συνεργάζονται στενά με την Κεντρική Τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ολλανδίας. Όμως, όσον αφορά την λειτουργία και ακαιρεότητα της Τράπεζας Κουρασάου Αγίου Μαρτίνου, η Τράπεζα οφείλει να επεκτείνει, η Κεντρική Τράπεζα δηλαδή, την εποπτεία της και στις χώρες αυτές. Επίσης, οι εισαγγελικές υπηρεσίες συνεργάζονται στενά και σε ζητήματα οικονομικού και φορολογικού χαρακτήρα. Το πολιτικό, νομικό και θεσμικό πλαίσιο των Μπονέα, Στάσια και Σάμπα είναι αρκετά απλό. Οι χώρες αυτές αποτελούν τμήμα των κάτω χωρών και επομένως η νομοθεσία τους για την φοροαποφυγή, ξέβλημα ε, μαύρου χρήματος και φοροαποφυγή θεσπίζονται από την Ολλανδική κυβέρνηση της Χάγης. Η εφαρμογή ε, γίνεται αντικείμενο εποπτείας από Ολλανδικούς θεσμούς, την Ολλανδική Κεντρική Τράπεζα καθώς και την Ολλανδική Αρχή Χρηματοπιστωτικών Αγορών. Έρχομαι τώρα στα βασικά μου συμπεράσματα. Όπως είπα, χρειάζεται μια πολυσχηδής προσέγγιση για να γίνει κατανοητό το πολυσχηδές θεσμικό πλαίσιο της Ολλανδίας. Σε ό,τι αφορά την χώρα της Ολλανδίας υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για την άσκηση επιρροής για την αντιμετώπιση τέτοιων δραστηριοτήτων στις ε, χώρες Μπονέα, Στάσια και Σάμπα που αποτελούν τμήμα της Ολλανδίας και ε, όπου βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Χάγης. Εκεί εφαρμόζεται η Ολλανδική νομοθεσία. και η επιβολή είναι επίση ζήτημα Ολλανδικό. Σε ό,τι αφορά τις τρεις αυτόνομες, σχεδόν ανεξάρτητες καραϊβικέ χώρε που ανήκουν στο βασίλειο της Ολλανδίας, οι δυνατότητε άσκησης επιρροή στον αγώνα κατά ε, της και κλπ. είναι μάλλον περιορισμένες. Στην Αρούμπα κλπ. έχουν καλώσει μεν στα χαρτιά, αλλά η εφαρμογή του νόμου είναι κάτι διαφορετικό στο επίπεδο του Βασιλείου οφείλουμε να συμπεράνουμε ότι η σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ολλανδίας και των καραϊβικών χωρών είναι αμφιλεγόμενη και ιδίω όσον αφορά τις αυτόνομες καραϊβικές χώρες Αρούμπα Κορασάου και Άγιο Μαρτίνο τοποθετούνται ανάμεσα σε ανεξαρτησία και εξάρτηση και σε αυτή την ενδιάμεση κατάσταση οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ολλανδίας κινούνται με πολύ μεγάλη προσοχή, οφείλω να πω. Είναι πολύ περιορισμένες οι τυπικές εξουσίες της Ολλανδικής κυβέρνησης. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν και αδυναμία επιβολής αντισταθμίζεται από συνεργασία, η οποία συχνά ξεκινά με πρωτοβουλία της Ολλανδικής Κυβέρνησης της Χάγης. Επομένως, στις καραϊβικές χώρες και όχι εδάφη, η διάκριση είναι ανάμεσα σε καραϊβικές χώρες και καραϊβικά εδάφη της Ολλανδίας, δεν είναι δεδομένη. Μπορεί να συμπληρώνεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί θα ληφθεί υπόψη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσα στα πλαίσια των υπερπόντιων ρυθμίσεων για τη λήψη αποφάσεων. Θα ήθελα να ολοκληρώσω με λίγες παρατηρήσεις σχετικά με το μέλλον του Βασιλείου της Ολλανδίας, που είναι πλήρες αβεβαιοτήτων και κινδύνων. Ιδίως η κατάσταση στην ε, Κουρασάου και στον Αγιο Μαρτίνο φαίνεται να είναι πολύ εύθραυστη. Ο μεγαλύτερος αριθμός των κατοίκων της Αρούμπα θέλουν να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ Αρούμπα και Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι η εντύπωσή μου, ο μεγαλύτερος αριθμός είναι υπέρ της ε, χορήγησης στη χώρα αυτή του καθεστώτος των υπερπόντιων εδαφών, ενώ στο Κουρασάο η κατάσταση είναι διαφορετική. Είναι μια πολύ μικρή πλειοψηφία αυτή που τάσεται υπέρ της συνεργασίας με το Βασίλειο και στο μέλλον μπορεί να αλλάξει, διότι υπάρχουν και ζητήματα διαφθοράς στον Άγιο Μαρτίνο πλέον, μπορεί ε, να αποτελέσει μοντέλο και για το βασίλειο της Ολλανδίας η γαλλική ε, θεσμική ρύθμιση, αλλά χρειάζεται να προσεγγίσει περισσότερο στην πολιτική πραγματικότητα. Συνεχίζεται πάντως το, η επεξεργασία του θέματος φόρα αποφυγής και της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών αυτού του Ατλαντικού. Μου εξήγησε η γραμματέα μου ότι δεν είναι γκρόνιγεν αλλά χρόνιγεν. Θα έπρεπε να τα καταφέρει καλύτερα γιατί κάποια Ολλανδικά είχα μάθει μικρό. Ζητώ συγγνώμη από του Ολλανδού. Και ο επόμενο είναι ο κ. Κλακ. Κλέγκ, συγγνώμη. Thank you very much. Uh, I just want to provide a brief... Να σας δώσω μια εικόνα του τι ισχύει για αυτές τις ε, υπερπόντιες ε, κτίσεις και περιοχές και εδάφη. <clears throat> Όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο, να σας πω ότι γίνεται όσον αφορά το νομικό καθεστώς και το πολιτικό καθεστώς που αφορά τις καθημερινές σχέσεις και επίσης επηρεάζει ε, τις οικονομικές και όχι μόνο σχέσεις. Και να δούμε επίσης ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο που διαμορφώνει την προσέγγιση μας και να σας πω και κάποια συμπεράσματα αλλά και συστάσεις. Πρώτα πρώτα για ρίξω μια ματιά ε, σε αυτά τα εδάφη. Τέσσερα είναι που έχουν σχέση με το Μέλλον Βασίλειο, έξι ε, αναφέρονται εδώ. Πάντως σε διαφορά με Γαλλία και κάτω χώρες η κάθε χώρα έχει διαφορετική ε, σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν ομοιότητες αλλά και ιδιαίτερε διαφορές ανάλογα με την ιστορία της κάθε χώρας, της κάθε περιοχής. Και πολλές φορές μία από τις κτήσεις ε, υπαγόταν σε μια άλλη, οπότε υπάρχει και διαφορετικό στεγματικό καθεστώς και αυτονομία που διέπει την καθεμία. Τέλος πάντων έχουμε κάποιο είδους βασικές ε, διατάξεις που διέπουν αυτές τις ε, σχέσεις και που προέρχονται και θεσπίζονται από το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά τις σχέσεις αυτές είναι επομένως από πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ε, βασικό όργανο το σύνταγμα που, του, συνταγματικού του χαρακτήρα διάταξη οπότε τουλάχιστον θεωρητικά ε, το δίκαιο του, Ηνωμένου Βασιλείου επ' αυτών των ε, περιοχών. Επίσης, όπως είπαμε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρα τα όρια της ε, κάθε εξουσίας και της ε, αυτονομίας και, και μάλιστα πρόσφατα έχουν χωριθεί περισσότερες εξουσίες και αυτονομία. Ε, υπάρχει γενικώ ε, οικονομική αυτάρχεια, υπάρχει ΑΕΠ αρκετά υψηλό, αλλά οι οικονομίες αυτών των περιοχών εξαρτώνται ε, από δύο βασικά θέματα. Είναι η θέμα βιωσιμότητάς τους δηλαδή. Όσον αφορά τώρα το τι ισχύει όσον αυτά τα τις οικονομίες, τη χρηματοοικονομική λειτουργία πλευρά νομική και πολιτική. Όλοι είπαν για τι τις Παρθένες το Virgin Islands και τα νησιά Cayman. Αλλά επίσης ε, αυτό αφορά και τη, τις βερμούδες τη από πλευρά ασφαλιών. Και έχουμε κάποιες διατάξεις από τη ΣΥΠΑ και έχουμε και κάποιο είδους ε, πρότυπα που έχει θεσπίσει ως το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει προσπαθήσει να συμβάλλει όσον αφορά τη σχετική ε, τραπεζική ε, οδηγία, τα, τελικά πίεσε το Ηνωμένο Βασίλειο και ίσχυσε αυτό το μέτρο και στα νησιά Κέιμαν. Και επίσης έχουμε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εδώ αλλά υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν επομένω κάποιου είδου ε, δομέ κανονιστικέ που είναι ενεπαρκεί. Είναι και θέμα ανθρωπίνων πόρων. Πολλέ φορέ λείπουν. Επίση, ε, πολλέ φορέ υπάρχουν σχετικέ υπηρεσίε δεν συμμορφώνονται με βασικά νομοθετήματα. Έχουμε επίση ε, πάρα πολύ λίγε καταδίκες σε αυτές τι περιοχές. Επίσης δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση για την πραγματική κυριότητα και υπάρχει νομοθεσία που απαγορεύει την καταγγελία και τη δράση πληροφοριδιωτών. Τώρα όσον αφορά την καθημερινή πολιτική λειτουργία, ε, Αγγίγια, Μοντσεράτ και Κάιμαν ε, εκεί ο κυβερνήτης ε, είναι ο πιο αρμόδιος για αυτούς τους τομείς και λογοδοτούν στο Λονδίνο εκπροσωπώντας ε, την περιοχή τους, τη χώρα τους. Επίσης εδώ όμως υπάρχουν κάποια σαφή θέματα είπαμε ότι λογοδοτεί στο Λονδίνο ο κυβερνήτης αλλά επίσης εκπροσωπεί και αυτή την κτήση. Αλλά είναι διπλός ο ρόλος τους και αυτό τους δυσκολεύει να μπορέσουν να καλύψουν και τα δύο μέτωπα. Να εκπροσωπούν δηλαδή τα συμφέροντα της χώρας και να λογοδοτούν και να ξέρουν ακριβώς και τι γίνεται. Τώρα είναι το θέμα του, της Υπάρχει αυτό το χρηματοδότηση θα μπορούσαμε να πούμε για κάθε τέτοια περιοχή έχουν προϋπολογισμό, μπορούν να αποφασίσουν τα δημοσιονομικά, τις δημόσιες δαπάνες και επίσης αποφασίζουν και για το τι ισχύει όσον αφορά τις εξωχώρες δραστηριότητε. Επίσης, ο κυβερνήτης προέρχεται από το Λονδίνο, αλλά δεν ξέρει αναγκαστικά την ε, περιοχή ή τη χώρα. Πρέπει να προσαρμοστεί θα πρέπει να μπει στα ενδότερα αυτών των πολλές φορές κλειστών κοινοτήτων. Αλλού δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο κυβερνήτης. Και έχουμε εκεί κάποιες επιτροπές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών όπως τα νησιά Καϊμάν. Εκεί υπάρχει συνεργασία, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εδώ μπορούμε να συγκρίνουμε τη σχήμη με τις κάτω χώρες δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη του Ηνωμένου τόσο ώστε να τους επιβάλλει να θεσπίσουν ένα πλαίσιο. Γνωρίζει το Ηνωμένο ότι υπάρχει βέβαια αυτή η αυτονομία και για αυτό δεν θέλει το Ηνωμένο να αναμειχθεί τι γίνεται σε κάθε μία από αυτές τις κτήσεις ή πρώην Πάμε πίσω στο 1989. Έχουμε την υπόθεση Σεράτη. Το 1989 είχε θεωρηθεί ότι γίνεται πάρα πολύ ξέβλημα χρήματος εκεί. Όμως η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη και ο κυβερνήτης ανέλαβε προσωπικά με τη βοήθεια της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να ελέγξει πάλι τα οικονομικά Έχουμε τελευταία το διάλογο που καλά κρατεί όσον αφορά τα θέματα και έτσι έχει, είναι δυνατόν, είπαμε, να έχουμε κάποιο είδους ε, καταλόγους, μητρώα για τους αληθείς κυρίως. Οπότε, να δούμε τώρα ποιο είναι το ευρύτερο πλαίσιο, η συγκυρία πολιτική και οικονομική Είπαμε τον Εμένο Βασίλειο διστάζει να χρησιμοποιήσει όλες τις εξουσίες που έχει. Πιστεύει ότι οι καλές σχέσεις με δημοκρατικές κυβερνήσεις είναι το πιο σημαντικό. Και πιστεύει η χώρα ότι θα πρέπει να ενθαρρύνει ε, αυτά τα εδάφη να αυτοδιοικούνται και να μην επιβάλλεται η κυβέρνηση από τα πάνω. Έχουν σημαντικέ δυνάμει εξουσία από το Σύνταγμα οι κυβερνήτε. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά το πράγματα στο προχώρητο, αλλά μπορούν επίση οι κυβερνήτε να χρησιμοποιήσουν τι εξουσίε του εκεί. Αλλά δεν μπορούν να έχουν τη διευκόλυνση κάποιων ενδιάμεσων για να ασκήσουν πιέσει. Κάτι το οποίο θα ήταν επιθυμητό και χρήσιμο. Επίσης, Δεν υπάρχει συνέχεια στο προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα θέματα από πλευράς κυβέρνησης της Αγγλίας. Υπάρχει δηλαδή η λεγόμενη συνταγματική θεσμική μνήμη. από πλευράς οικονομικής συγκυρίας. Δεν νούμερο βασιλό αποφασισμένο να προσδώσει αυτάρκεια οικονομική στη ε, εδάφια αυτά. Οπότε είναι πολύ σημαντικά και κάθε επιδείνωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση της στήριξης από νόμο Βασίλειο, κάτι που δεν το θέλει το νόμο Βασίλειο. Επίσης, θεωρούν αυτά τα εδάφη και εκτίσεις ότι η αυτονομία οδηγεί και στην πολιτική αυτονομία. Άρα θέλουν να μπορούν να στέκονται στα πόδια τους όσον αφορά τα οικονομικά και την ανάπτυξή τους. Επίσης για τα οικονομικά βεβαίως και υπάρχουν ισχυροί δεσμοί με το ΣΥΤΙ και αυτού του είδους τα εξωχώρια κέντρα. Ωραίες σημαντικές μεταξύ του ΣΥΤΙ και αυτών των περιεχών. Τέλος, ο πρόεδρος οικονομικής από την κρίση του 2007-2008 προσπάθησε κάπως να κρατήσει τα ηνία το Ηνωμένο Βασίλειο, να σφίξει τα λουριά και τελικά όμως και πέραν της κρίσης συνέχισε να ισχύει η πεποίθηση ότι πρέπει να έχουν αυτονομία οικονομική οι περιοχές αυτές. Βέβαια ενθαρρύνονται οι περιοχές αυτές να έχουν πιο υγιεινή μισονομικά και όταν σε πολλές περιοχές υπήρξε μεγάλη δυσκολία, το 2008-2009 η εργατική κυβέρνηση είπε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο είδους φορολογία για τα νησιά Κέιμαν. Αυτό ήταν μια πρόταση όμως που μπήκε στο ψυγείο όταν έπεσε η κυβέρνηση των εργατικών. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό το τι θα γίνει τα αυτά τα εξωχώρια χρηματοοικονομικά, ε, και οι περικοπές των δαπανών ε, και καλύτερη νομοθεσία θα βοηθούσε. Οπότε θέλουν να διατηρηθεί αυτή η εξωχώρια δραστηριότητα γιατί είναι σημαντική για την οικονομική υγεία των χρόνων αυτών. Τώρα, σαν συμπεράσματα και συστάσεις, είπαμε ότι είναι κυρίαρχο το Ηνωμένο Βασίλειο και ε, τελικά κατησχύει ε, αυτών των τοπικών κυβερνήσεων έχουν πάντως μεγάλη αυτονομία ε, αυτά τα εδάφη, αλλά βέβαια ε, τελικά ε, αυτό το θεωρητικό πλαίσιο δεν ισχύει αναγκαστικά και πολλές φορές δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία όπως και όποτε και όσο πρέπει τοπική αυτονομία κατησχύει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει συνεργασία ούτως ώστε να πλαισιωθεί ο τομέα των χρηματοοικονομικών, θα αυτό επιδέχεται βελτίωση. Πρώτα-πρώτα θέλουμε περισσότεροι πόροι να βοηθήσουν ναι, να, να, να συντελέσουν σε καλύτερο πλαίσιο. Αγωνιστικό. Επίσης θα πρέπει να δούμε πέραν των χρηματοοικονομικών τι γίνεται, να υπάρχει περισσότερη ισορροπία στην οικονομία και το νομένο Βασίλειο να έχει πιο αποφασιστικό ρόλο και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και πώς η τοπική ανάπτυξη θα συνδεθεί περισσότερο με τις χρηματοοικονομικές εξωχωρές δραστηριότητε. Και μία θα βοηθήσει την άλλη. Συνεχίζουμε και βοηθούμε αυτά τα εδάφη. Αλλά βέβαια αυτό που χαλάει τη συνταγή είναι το Brexit. Το Brexit θα επιδεινώσει τα πράγματα. Και δεν θα βοηθήσει όσον αφορά το πώς αυτά τα εδάφη θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα λόγω προβλήματα. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταία παρουσίαση, παρουσίαση είναι η περίπτωση της Γαλλίας, των γαλλικών περπόντιων ε, εδαφών και χωρών. Αλεξάνδρα Μετρόντε Λαμότ είναι ομιλητής που θα μας μιλήσει στα γαλλικά. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι πολύ που μπορώ σήμερα να σας παρουσιάσω την έγγραφη εργασία μου ε, των τελευταίων μηνών. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Προκατακτικά ευχαριστώ τις ε, υπηρεσίες μου, τα μέλη του Exposed Evaluation Unit και βλέπετε τα ονόματά τους. Εδώ βλέπετε τα τέσσερα, τα πέντε συγγνώμη εδάφη στη διαφάνεια. Εξελίσσονται τα πράγματα βέβαια θεσμικά. Μετά θα δείτε και το χάρτη. Βλέπετε τα Σεντ Μπαρτελέμι, Σεντ Πιέρ Μικελό, Σεντ Φουτούνα και η Γαλλική Πολυνησία και η Νέα Καλλιδονία. Το αρχιπέλαγος αυτό με τις τέσσερις αυτές, με τα τέσσερα αυτά εδάφη και υπάρχουν και άλλα υποσύνολα βέβαια. Ποια είναι η εξέλιξη. Σαν παρτελεμία αρχικά, στην πρώτη δηλαδή ε, συνθήκη της, ε, για τη λειτουργία της Ένωσης δεν συγκαταλεγόταν ε, στα γαλλικά είχε. Ήταν η Γουαδελούπη, μετά ξεχωρίστηκε το Σαν Παρτελεμή και αποτελεί ξεχωριστό είχε. Και σε αυτό τον κατάλογο θα βρείτε και τη Μαγιότ, που όμως στο μεταξύ έχει γίνει υπερπόντε διαμέρισμα. Α, ορίστε και ο χάρτης που σας έλεγα. Δείχνει γεωγραφικά πώς ε, κατανέμονται αυτές οι υπερπόντες χώρες και εδάφη. Στο 73 και 74 του συντάγματος της Γαλλίας έχουν ε, το καθεστώς της συλλογικότητας, κολεκτιβιτέ, λοκάλε τεριτοριάλ αυτά τα εδάφη. Βέβαια είναι πολύπλοκα τα πράγματα. Έχουμε τα διαμερίσματα και τις περιφέρειες, ε, Μαρτινίκα, Γουαδελούπη και Γαλλική Γουιάννα, στον Ατλαντικό και στον Ινδικό. Από το 2014 έχουμε τη Μαγιώτα που πριν ήταν ε, ΠΤΟΕΜ, και τη Ρενιόν. Μετά έχουμε τις υπερπόντιες συλλογικότητες, κολεκτιβιτέ ντούτρ με άλλο καθεστώς από το καθεστώς του διαμερίσματος που ήταν τα πρώτα με τον μπλε που σας έδειξα. Είναι όμως υπερπόντιες χώρες η εδάφη, βλέπετε στον Ατλαντικό το Σεμπιέρε Μικελόν, το Σεν και το Σεμπαρτέλεμι. Το Σεμαρτέν δεν είναι όμως υπερπόντια χώρα ή έδαφος σύμφωνα με το δίκαιο, αλλά ε, είναι αξιόχως απόκεντρη η περιφέρεια, ενώ το Σαν που αρχικά ήταν υποσύνολο του, διαμερίσματος, του υπερπόντιου διαμερίσματος, που ήταν και εγώ τώρα έχει γίνει ε, χώρα, υπερπόντιο έδαφος και περιλαμβάνεται στη μελέτη μας ως κολεκτιβιτέ ντουτρμέρ. Έπειτα βλέπουμε τρία ε, συμπλέγματα νήσων. Ε, έχουμε τη Γαλλική Πολυνησία, Γόλης και Φουτούνα και Νέα Καλυδονία. Υπάρχει μια κάποια αντιστοιχία μεταξύ αυτών που προβλέπει το Γαλλικό Συνταγματικό Δίκαιο αφενός ε, και το Δίκαιο της Ένωσης αφετέρου. Με το κόκκινο σε αυτό το συγκεφαλαιωτικό πίνακα βλέπετε τις συλλογικότητες, αυτούς, αυτές τις περιοχές που τις θεωρούμε άκρος απόκεντρες περιφέρειες και δεν τις μελετούμε, για τον πολύ απλό λόγο στην προκειμένη περίπτωση ότι το πρωτογενές δίκαιο και το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εφαρμόζονται αυτομάτως και άμεσα ο Γάλλος νομοθέτης κάθε φορά που μεταφέρει μια ευρωπαϊκή οδηγία για παράδειγμα θα πρέπει να καλύψει και αυτά τα εδάφη γεωγραφικά. Μας ενδιαφέρουν λοιπόν τα εδάφη τα οποία είναι με λευκό στην ε, αριστερή στήλη, το Σεν Παρτελεμή, το Σεν Πιέρε Μικελόν, το Γόλις και Φουτούνα, η Γαλλική Πολυνησία και η Νέα Καλυδονία. Θα πρέπει να ξέρετε επίσης ότι σύμφωνα με το Γαλλικό Συνταγματικό Δίκαιο υπάρχουν δύο νομικά καθεστώτα που εφαρμόζονται ε, τα βλέπουμε στο μέσο ε, με το COM, Collectivité d'Outre-mer. Έχουμε το AS που σημαίνει assimilation, αφομοίωση, το SP που σημαίνει specialization, εξειδίκευση. Με διαφορετικές μεθόδους ουσιαστικά στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγουμε. Όταν εφαρμόζεται το καθεστώ τη αφομοίωση ασημιλασιών, τι ισχύει. Οι γαλλικοί, οι μετροπολιτικοί νόμοι εφαρμόζονται εκτό ε, αν προβλέπουν κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, Ισχύει το πολιτικό δίκαιο, εκτός αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, παραδείγματος χάρη αν έχουμε διαφορετικές διατάξεις, φορολογικά θέματα για το επίπεδο των φόρων, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Παραδείγματος χάρη διοικητική συνεργασία, ξέπλυμα χρήματος κτλ. Στο άλλο καθεστώς τώρα, σπεσιαλιζασιό, εξειδίκευση, εδώ έχουμε μια άλλη λογική, η οποία εφαρμόζεται και στο πλαίσιο της μελέτης μας βέβαια καταλήγει στο ίδιο αποτέλεσμα. Η αρχή είναι ότι το πολιτικό δίκαιο εφαρμόζεται μόνο αν το γαλλικό Κοινοβούλιο, η Γαλλική Βουλή ε, το αποφασίζει. Αν δηλαδή αποφασίσει ότι θα επεκτείνει και σε αυτά τα εδάφη ε, τη γαλλική νομοθεσία το Κοινοβούλιο, τότε θα ισχύσουν οι διατάξεις, ε, παραδείγματο χάρη για τους φόρους. Αφήνει πάρα πολύ μεγάλο περιθώριο στις συγκεκριμένες περιφέρειες το Κοινοβούλιο. Αλλά σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση του ξεπλήματο χρήματο ή την, οργασία, την οργάνωση διοικητική συνεργασία, ο Γάλλο νομοθέτη επιλέγει πάντοτε να προβλέψει την ε, επέκταση ε, τη ισχύω ε, του γαλλικού δικαίου σε αυτέ αυτές τι περιφέρειε, σε αυτά τα εδάφη. Το αποτέλεσμα βέβαια για τη δική μα τη μελέτη πάντοτε είναι το ίδιο. Υπάρχει κάποια αυτονομία αυτών των περιοχών για φορολογικά θέματα, για τη φορολογική βάση, για του κανόνε σύσπραξη κτλ. Όμως εφαρμόζεται είτε στην περίπτωση της αφομοίωσης είτε στην περίπτωση της εξειδίκευσης στο μητροπολιτικό δίκαιο σε αυτές τις υπερπόντες χώρες και εδάφη μας ενδιαφέρουν στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος ή στα θέματα διοικητικής συνεργασίας διότι ο νομοθέτης, ο Γάλλος νομοθέτης έτσι θέλησε. Γενικά τώρα πρέπει να δούμε ότι αυτές οι υπερπόντιες συλλογικότητες, τα υπερπόντια αυτά εδάφη, ε, δεν έχουν κυριαρχία και έχουν κάποιες αρμοδιότητες που προβλέπει το Σύνταγμα. Δηλαδή το Σύνταγμα και η εθνική νομοθεσία αποφασίζουν τι δικαιώματα έχουν και τι δεν έχουν αυτά τα εδάφη Υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία έχουν αυτονομία και κάποια όχι. Μπορεί να του χωρί κάποιε αρμοδιότητε, ε, δηλαδή η Μητροπολιτική Γαλλία, αλλά μπορεί και να του αφαιρέσει ανα πάσα στιγμή. Και στην προκειμένη περίπτωση μα ενδιαφέρει, επαναλαμβάνω, υπάρχει κάποια αυτονομία για τα φορολογικά ζητήματα, καμία όμω αυτονομία δεν εκχωρείται για την καταπολέμηση του ε, ξεπλήματο ε, χρήματο και σε θέματα διοικητική συνεργασία. Εδώ έχετε κάποια αριθμητικά στοιχεία για πληθυσμό, ΑΕΠ και κάποιου βασικού τομεί. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, οικονομικής φύσης πρέπει να έχετε υπόψη είναι ότι ε, αυτά τα γαλλικά υπερπόντια, αυτές οι κτήσεις ε, είναι σχετικά φτωχές. Βλέπετε τι ισχύει για ορισμένε περιπτώσεις. Οι ενισχύσεις που δίνει η Μητροπολιτική Γαλλία, ε, οι οικονομικές ενισχύσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές. Αν δείτε τη γαλλική πολυνησία Νέα Καλλιδόνια, τα δύο τελευταία δηλαδή, βλέπετε ότι ξεπερνάμε το δις, τον, το δις ευρώ οικονομικής ενίσχυσης ε, ετησίως για την κάθε μία ε, αυτή περιοχή. Και ο δημόσιος τομέας είναι συνήθως ο βασικότερος τομέας δραστηριότητας που όπως είπαμε χρηματοδοτείται από το Μητροπολιτικό ε, κράτος. Εδώ τρία βασικά σημεία, φοροαποφυγή, καταπολέμηση ξεπλήματος χρήματος και δημοσιονομική φορολογική διαφάνεια. Θα σας πω επίσης σε κάθε περίπτωση ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσαμε. Πρώτα απ' όλα, φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή. Εδώ ε, κάτι που μας ενοχλεί ιδιαίτερα και μας προξενεί ενόχληση είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε να βρούμε στοιχεία. Είναι πάρα πολύ λίγα, πολλές φορές είναι απαρχιωμένα. Ε, αν διαβάσετε την έγγραφη έκδοση έκθεση θα δείτε ότι φτάνουμε στο 2010, 11, το πολύ, ε, που σημαίνει ότι δεν παράγονται δεδομένα από τις τοπικές αρχές και το ελεγκτικό συνέδριο εκφράζει πολλές φορές παράπονα για αυτή την κατάσταση, αλλά και άλλοι φορείς ε, ελέγχου εκφράζουν παράπονα και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Έχουμε ένα πρόβλημα με τα slides. Εσείς συνεχίστε, Πρέπει να δούμε εδώ αν υπάρχει κίνδυνος φόρο διαφυγής από αυτά τα υπερπόντια εδάφη χώρες. Ε, πώς έχει κατάσταση. Εδώ ε, υπάρχουν διαφορές, ε, ποικίλη κατάσταση. Εκεί που μπορεί να υπάρχει πρόβλημα είναι όταν είναι λίγη η άμεση φόροι. Στο ΣΕΠΑΡ αυτό το επέλεξε η ίδια αυτή η περιφέρεια, δεν υπάρχει φόρος εταιριών ή φόρος επί του εισοδήματος άλλο για τους ε, νέους πολιτογραφηθέντες πάλι, αλλά υπηκός, αλλά για τους ε, υπηκός ε, του Σαν Παρτελεμή δεν ισχύει. Για Γαλλική Πολυνησία και την Καλιβωνία και το Σαν Μικρό, σε ό,τι αφορά τις κατώτατες πράξεις φόρων, είναι λίγο πολύ το επίπεδο αντίστοιχο με το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν έχουμε ασθενή φορολόγηση είτε για τη βάση είτε για τους συντελεστές. Μια άλλη δυσκολία εδώ που αντιμετωπίζεται ότι επειδή δεν υπάρχουν μέσα, οι φορολογικέ ε, διοικήσει που δεν έχουν ε, μέσα στη διάθεσή του δεν μπορούν να ελέγξουν επαρκώ τα πράγματα ε, και δίνω κάποια στοιχεία στην έρευνά μου που δείχνουν ότι είναι πολύ λίγοι πόροι αυτοί και γι' αυτό και τα αποτελέσματα είναι περιορισμένα σε ό,τι αφορά τους ελέγχους. Επομένως αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε διαθέσιμα στοιχεία. Βέβαια όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια προοπτική και να μην υπερβάλλουμε Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πω ότι η φορολογία είναι πολύ ευνοϊκή για τους κατοίκους, αλλά πάρα πολύ ε, ε, τιμωτική για τους ε, ε, ε, ξένους. Για το Σεν Παρτελεμή, πριν πάρει κανείς το καθεστώς του φορολογικού υπηκόπου, περάσουν πέντε χρόνια Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι γεωγραφικές αποστάσεις και δυσκολία πρόσβασης. 24 ώρες και παραπάνω χρειάζεται να πάει κανείς από το Παρίσι στη Γαλλική Πολυνησία και σε ό,τι αφορά το ξέπλυμα χρήματος έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Το τραπεζικό σύστημα επιτόπου είναι πρωτόγωνο θα έλεγα κατά κάποιο τρόπο και επομένως δεν επιτρέπει την ε, πραγματοποίηση σοφιστικέ συναλλαγών. Πάμε στο θέμα του ξεπλήματος χρήματος. Εδώ πρέπει να ξέρετε ότι παραδοσιακά ο Γάλλος νομοθέτης πάντοτε επιλέγει να εφαρμόσει σε αυτά τα εδάφη και χώρε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δηλαδή κάθε φορά που πρέπει να μεταφερθεί μια ευρωπαϊκή οδηγία στο εθνικό δίκαιο, ο Γάλλος νομοθέτη δεν υποχρεούται μεν, αποφασίζει όμω ε, να επεκτείνει του κανόνε αυτού, ε, να εφαρμόζονται δηλαδή και στι ε, υπερπόντε χώρε και εδάφη και όταν υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κανονισμό, η επιλογή που γίνεται είναι να μεταφέρονται αυτομάτως αυτές οι διατάξεις και να ισχύουν και στα ΙΧΕ. Αυτό είναι η κλασική κατάσταση. Αν να δούμε τον τελευταίο κανονισμό, την τελευταία οδηγία, θα δείτε ότι το Δεκέμβριο του 2016 εγκρίνεται αυτή η σχετική νομοθεσία και εφαρμόζεται και στα ε, υπερπόντια εδάφη και χώρες. Βέβαια υπάρχει μια διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης πάλι σε ό,τι αφορά τη δήλωση υποψίας όπως το λέμε, reporting of suspicions. Υπάρχει ε, ανεπάρκεια οι συμβολιογράφοι, τράπεζε θα πρέπει να απευθύνουν αυτές τις ε, εκθέσεις. Δεν ξέρετε, δεν γίνεται όμως αυτό που θα έπρεπε να γίνεται στα υπερπόντα εδάφη σε σχέση με το ότι γίνεται στην Μητροπολιτική Γαλλία. Και πάρα πολύ λίγοι έλεγχοι επίσης γίνονται από τη στιγμή που έχουμε και πολύ μικρό reporting of suspicion στην αρχή. Και μια άλλη δυσκολία είναι η έλλειψη δεδομένων δεν υπάρχει, αν θέλετε, κουλτούρα για την καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος ε, από τους τοπικούς επαγγελματίες. Εδώ βέβαια έχουμε και ένα άλλο θέμα. Πώς, αφού μας ενδιαφέρει ε, το τραπεζικό σύστημα, βλέπουμε ότι ναι μεν είναι οι κίνδυνοι περιορισμένοι, έχουμε θηγατρικές γαλλικών ομίλων και όχι άλλα τραπεζικά ιδρύματα και μάλιστα πολλά είναι θηγατρικές δημόσιων ιδρυμάτων. Άρα έχουμε κίνδυνους, μικρούς κινδύνους. Εγώ εξέτασα τον αριθμό των τραπεζικών λογαριασμών και τι ποσά περιλαμβάνουν, γιατί υπάρχει μια κεντρική βάση της Τράπεζας της Γαλλίας ή το Institut de Mission Monetaire από τα υπερπόντια εδάφη στη Γόλη και το 70% του πληθυσμού μάλιστα δεν είχε καν ε, λογαριασμό στην τράπεζα. Έρχομαι στο τελευταίο που είναι η φορολογική διαφάνεια. Υπάρχει δυνατότητα ανταλλαγή πληροφοριών, υπάρχουν σχετικές συμφωνίες, βλέπετε τις διατάξεις. Η Γαλλία γενικά πρέπει να πω ότι υπερβαίνει τα πρότυπα του ΩΣΑ μπορεί η Μητροπολιτική Γαλλία να ασκεί φορολογικούς ελέγχους ε, στα ΙΧΕ ή να κοινοποιεί πάρα πολύ εύκολα ε, και να λαμβάνει πληροφορίες. Πάλι όμως μας ε, ενόχλησε το γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή δεδομένα. Στην έκθεση του ΟΣΑ του 13 εδώ παρόλα αυτά λέγεται ότι είναι υποδεγματική η Γαλλία παρόλα αυτά ε, η Γαλλία λέει ότι υπάρχει κίνδυνος ασυμμετρίας, ε, ότι εμείς ε, συνεργαζόμαστε υπερβολικά και άλλοι συνεργάζονται πάρα πολύ λίγο. Τέλος πάντων, πολύ λίγοι είναι οι κίνδυνοι, θεωρητικά ή πρακτικά για τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της κατάστασης που υπάρχει στα υπερπόντια εδάφη και χώρες. Τρεις παράγοντες βλέπουμε εδώ. Τον έλεγχο του κεντρικού κράτους, πρώτος παράγοντας. Δεύτερον, ότι εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ακόμη και αν δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση. Και τρίτον, βλέπουμε ότι γενικότερα ούτε οι οικονομικές δομές, ούτε οι τραπεζικές δομές ουσιαστικά ευνοούν αυτές τις πρακτικές που είναι κατακριτές και καταδικαστές. Σίγουρα υπάρχουν περιθώρια βελτιώσεων, μια καλύτερη κουλτούρα, περισσότεροι πόροι, περισσότερη ευαισθητοποίηση στους κινδύνους και ποια είναι, ποιο είναι το συμπέρασμα το τελικό. Ε, αν το γαλλικό μοντέλο μπορεί να είναι ένα μοντέλο και για άλλους, ε, αυτό είναι το ερώτημα, το είπαν και νομίζω οι δύο προλαλήσαντες, οι συγητές. Ίσως θεωρητικά είναι ωραία αυτή η φιλοδοξία, αλλά στην πράξη νομίζω είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Ευχαριστώ. Ε, merci beaucoup ε, Πρόεδρος Ντεμπάζη, σας ευχαριστώ και ευχαριστώ που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν είναι εύκολο, γιατί έχετε και πολλές πληροφορίες που επιθυμείτε να μας δώσετε. Ελπίζω ότι τα μέλη μας επωφελήθηκαν από αυτό μάθημα γεωγραφίας. Εγώ πάντως πολύ το απίλαυσα. Και ας περάσουμε τώρα στον πρώτο ομιλητή, που είναι ο συνεισηγητής της Επιτροπής Πάνα, ο κ. Κόφοντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος, γιατί δεν έχουμε πια πολύ χρόνο. Σας ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις σας. Πρώτα θα ήθελα να πω ότι αυτό που εξετάζουμε και στην Επιτροπή μας εδώ είναι η διασύνδεση μεταξύ ενδιαμέσων και κέντρων offshore. Και τα υπερπόντια αυτά διαμερίσματα είναι πολύ σημαντικά για μας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε από την έρευνα που κάνατε. Βλέπετε κάποιους βασικούς δείκτες που μπορούν να καθορίσουν ποιος είναι ο φορολογικός παράδεισος. Δεύτερο, ποια θα ήταν τα βέλτιστα κριτήρια για τους φορολογικούς παραδείσους από την άψη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τρίτο, για την ομοθεσία, εφαρμογή και επιβολή τα πρότυπα που έχουμε διεθνώς πρότυπα διαφάνειας κλπ. Ο ΣΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς τα βλέπετε να εφαρμόζονται με περισσότερο αποτελεσματικό τρόπο, άμεσα στα υπερπόντια αυτά εδάφη. Ή αρκεί οι ευρωπαϊκές χώρες με επίπεδο διαθέτουν τα εδάφη αυτά να προωθήσουν την εφαρμογή των συμφωνημένων αυτών προτύπων. Ας προσπαθήσει ο κάθε ομιλητής να απαντήσει στο ερώτημα αυτό ε, έχοντας διαθέσει τον λεπτό. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Οι βασικοί δείκτες, αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, για φορολογικούς παραδείσους, οι χώρες του Βασιλείου της Ολλανδίας όπως βρήκαμε εμείς στη μελέτη μας δεν είναι πολύ σημαντικές. Διότι η, βασική του, η βασική τους τομής οικονομικής δραστηριότητας είναι ο τουρισμός. Άλλωστε θυμηθείτε ότι είναι πολύ μικρά νησιά. Η Στάσια και η Μπονέρ, έχει, η Μπονέρ έχει 17.000 κατοίκους. Στάσια και Σάμπα έχουν 1.500 με 2.000 και η Σάμπα έχει μόνο 500 κατοίκους και ένα σχολείο. Η οικονομία λοιπόν συνδέεται πολύ στενά με τον τουρισμό, με μεγάλα διεθνή ξενοδοχεία, που αυτά εφαρμόζουν διεθνή πρότυπα στις δραστηριότητές τους. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ο τομέας φορολογικού παραδείσου και νομοποίησης παράνομων κερδών. Τώρα ποια θα ήταν τα βέλτιστα κριτήρια. Η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Η νομοθεσία της Σάμπια είδαμε σήμερα ότι είναι δύσκολη η εφαρμογή αφού περιλαμβάνει πολλές ασαφείς έννοιες ανοίγεται ένα πεδίο εφαρμογής του ατελούς δικαίου που δεν προβλέπει κυρώσεις δηλαδή και αυτό σημαίνει κατά τη γνώμη μου ότι η διαφάνεια εκεί μπορεί να αποδειχθεί προβληματική για την τρίτη σας ερώτηση το είδος της νομοθεσίας το είδος της ρύθμισης και πώς μπορεί να βελτιωθεί το, το επίπεδο εφαρμογής. Αυτό όντως είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Εκτός της επικράτειας του Βασιλείου Ολλανδίας όπως εξήγησα η Ολλανδική διοίκηση, εκτός αυτής δηλαδή, αλλά ομιλώντας για τις τρεις αυτές χώρες, κτίσεις δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει δυνατότητα άσκησης εξουσίας του βασιλείου της Ολλανδίας και επομένως ούτε της χώρας της Ολλανδίας, ας το πω, της Ευρωπαϊκής δηλαδή. Διακόπτει ο Ντεμπάζη, επειδή υπάρχει κάποιος περιορισμός χρόνου. Ας συμπλώσουν οι δύο άλλοι ομιλητές. Δεν διαφωνώ με τον συναδελφό μου, λέει ο κ. Κλέγκ. Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που βλέπετε όταν επισκέπτεστε τα υπερπόντια εδάφη είναι το ενδιαφέρον που έχουν για τους οικονομικούς τομείς σε σύγκριση με το μέγεθος και τον πληθυσμό τους. Μίλησα για την καπάστη, για την ικανότητα. Δηλαδή, είναι έτοιμη να εφαρμοστεί νομοθεσία αλλά το ερώτημα είναι αν υπάρχει ικανότητα επιβολής της. Και πάλι η φύση αυτών των μικρών κοινωνιών όπου όλοι γνωρίζουν όλους και αν έχει κανείς την αυτοπεποίθηση να βγει και να μιλήσει, να καταγγείλει δηλαδή πράγματα που μπορεί να συμβαίνουν. Και τέλος ό,τι αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα υπερπονδία εδάφη νομίζω ότι ήταν ε, σημαντικό πλήγμα η Βρετανική έξοδος θα ήθελαν να έχουν φωνή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούν να μιλούν για τα πράγματα αυτά και να είναι εντός όταν διαμορφώνονται οι πολιτικές που τα αφορούν. Πρώτα για τους βασικούς δείκτες που επιτρέπουν να χαρακτήσει ένας φορολογικός παράδεισος. Πρώτος Πρώτο, το επίπεδο της επιβολής, επιβολής δηλαδή το επίπεδο των φόρων που πληρώνεται εάν μια επιχείρηση δρά στην επικράτεια αυτή ή σε μια άλλη επικράτεια. Άλλος δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι το ζήτημα της συνεργασίας των διοικήσεων. Δηλαδή, εάν μια φορολογική διοίκηση μιας χώρας μέλους ζητεί προφορίες για μια επιχείρηση για έναν φορολογούμενο που βρίσκεται σε άλλο έδαφος, σε άλλο υπερπόνητο έδαφος, είναι θετική, αντική η στάση της άλλης διοίκησης και επαρκής ή όχι. Αυτό που συμβαίνει στα πλαίσια του ΩΣΑ, της peer review, της, ε, του ελέγχου των ομοτήμων δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και απέναντι σε χώρες που δεν συνεργάζονται. Το <coughs> επίπεδο επιβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο, γιατί είναι μάλλον ποσοτικό. Πρώτο κριτήριο, πόσες εταιρείε υπάρχουν ανά κάτοικο. πού ευρίσκεται ένα έδαφος, ένα υπερπόντιο έδαφος για παράδειγμα, σε σύγκριση με τον μέσον όρο όσον αφορά την, ε, τον αριθμό εταιριών ανά κάτοικο. Το ίδιο ο αριθμός τραπεζικών λογαριασμών που ανοίγονται σε μια χώρα, καθώς και το τι αποδίδουν για το ε, ΑΕΠ του συγκεκριμένου αυτού εδάφους. Όσο περισσότερα, τόσο μεγαλύτερο είναι ο κίνδυνος. Τέλος, ζήτημα της νομοθεσίας και της εφαρμογής της. Διακόπτει ο πρόεδρος δεν βάζει. Λυπούμε πολύ αλλά είμαστε υποχρεωμένοι. Δεν φταίτε εσείς. Δυστυχώς είναι η διαχείριση του χρόνου που έχουμε κάνει. Πρέπει να προχωρήσουμε λίγο. Σας παρακαλώ να συντομεύσετε λοιπόν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ζητήσει να δοθούν περισσότερες δυνατότητες στις χώρες μέλη να βλέπουν πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία. Ο συνηγητής της ομάδας Άλντε δεν είναι παρόν, άρα μπορούμε να προχωρήσουμε στον κύριο Νίτερ Μάιερ του Λαϊκού Κόμματος. Πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Για να δούμε. Είπατε, θέλουμε είπατε ότι είναι πάρα πολύ αυστηρή η ρύθμιση για του εξωτερικών χρημάτων και λοιπά στον Βασίλειο. Οπότε το πνεύμα που διέπει την νομοθεσία για τα Virgin Islands είναι αυτό. Και όταν συζητήσαμε εδώ με τους εκπροσώπους τραπεζών μας είπαν ότι στα εδάφια αυτά ισχύουν ακριβώς τα ίδια πρότυπα για τον εντοπισμό των πραγματικών κυρίων κλπ. κλπ. Ισχύει κάτι τέτοιο. Τι λέτε. Υπάρχουν πολλέ τράπεζε και λειτουργούν που δεν υπάγονται στους τραπεζικούς ομίλους, του ευρωπαϊκούς. Οπότε αυτό με προβληματίζει. Ποιον ωφελεί αυτό, εκτός βέβαια από αυτούς που εμπλέκονται εκεί. και είναι φυσικά μεγάλο ποσοστό των ασχολουμένων με αυτές τις εξωχώρες δραστηριότητες. Τι γίνεται, δεν χρειάζονται δημοσιονομικές ροές τα νησιά από την ενδοχώρα, την μητέρα χώρα. Κύριος Κλέγκ. Αυτό αντιστοιχεί στα όσα θα ήθελε το Ευρωπαϊκό να ισχύει και μέσα στη χώρα. Αλλά υπάρχουν κάποιε διαφορέ σε προσέγγιση, χρηματοδότηση, εφαρμογή. Πολύ σημαντικό επίση το ότι πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει αυτονομία σε αυτά τα εδάφη. Δεν θέλουμε να του βλέπουμε ω απικία μα πλέον. Οπότε δεν έχετε επίση παρά σε πολύ συγκεκριμένε περιπτώσει. Και όπω είπατε, έχετε δίκιο. ότι είναι θέμα μισονομικής ενίσχυσης σαν προσδοκία που ισχύει και κάτι το οποίο είναι ριζωμένο αυτό στην αντίληψη για το, τη σχέση που έχουμε με τα εδάφια αυτά. Οπότε άπαξ και υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι αποδεκτό, έτσι γίνεται. Αλλά σε την περίπτωση θα πρέπει να πάρει την θέση του. Γιατί πολλές φορές τα συστήματα αυτά, τα σχήματα αυτά υπάρχουν εδώ και μια σαρανταετία, ε, οπότε είναι ριζωμένα εκεί. Και άρα θέλει χρόνο ούτως ώστε κάποιος να φέρει την αλλαγή στο μοντέλο ανάπτυξη. Και θέμα είναι να υπάρχει οικονομική δυνατότητα και πολιτική βούληση να γίνει κάτι τέτοιο αποτελεσματικά. Κάποιος να συμπληρώσει, όχι. Πολύ ωραία λέει ο Πρόεδρος και προχωρούμε. Δεν θέλει άλλο το λόγο. Χωάν Φερνάντο Λόμπες Αγγιλάρ από την Σοσιαλδημοκρατική Ομάδα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές. Πιέζει ο χρόνος οπότε να προσπαθήσω και εγώ να εστιαστώ το τι γίνεται με τις υπερπόντιες κτίσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και λέμε στο παράδειγμα 2 της Συνδίκης της Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί έχουμε ένα μεγάλο νομικό πρόβλημα και πρόκληση. Όσον αφορά το να καταφέρουμε να καταπολεμήσουμε τις πρακτικές αυτές, τη φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα, διαπιστώσαμε ότι κάπως το γαλλικό μοντέλο ισχύει και εφαρμόζεται όσον αφορά την εφαρμογή και υλοποίηση των βρετανικών προτύπων. Οι δε ολλανδικές κτήσεις έχουν κάνει ένα βήμα παραπάνω, αλλά το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτές οι βρετανικές πρώην κτήσεις. Και ιδίω τώρα που έχει ανακοινωθεί η αποχώρηση, το Brexit. Κατά τη δεν υπάρχει νομικός τρόπος να εξασφαλίσουμε την ε, εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου για τα προβλήματα αυτά, Δηλαδή φορολογική διαφάνεια, δηλαδή ξέπλυμα, φοροδιαφυγή. Επομένω, εδώ ε, εγκυμονείται μια πραγματική απειλή του να υπάρχει παραθυράκι στο κοινωνικό δίκαιο. Οπότε, για πέστε μου, υπάρχει κάτι στο κοινωνικό δίκαιο, ούτως ώστε να ισχύει δεσμευτικά για αυτά τα εδάφια και τα εδάφια που θα μείνουν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση. που θα μείνουν τα κράτη-μέλη. Και επίση έχουμε τώρα αυτό το παραθυράκι, αυτό το νομικό κενό που διαπιστώθηκε. Ποιε είναι οι συνέπειε του Brexit για την εφαρμογή του Βρετανικού Δικαίου. Υπάρχει προβλέψιμη συνέπεια για το τι θα γίνει σε αυτά τα εδάφια ακριβώς λόγω του Brexit. Να δούμε και πώς θα οι εργασίες της Επιτροπής μας για το πώς τελικά θα προταθεί και θα, θα, θα καταλήξουμε σε κάποιο είδους κοινωτικό δίκαιο για τις χώρες που θα μείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή τις κτήσεις της Ολλανδικές και της Γαλλικές. Όλα αυτά τα χρήματα που πάνε εκεί πέρα, τι θα γίνει. Μήπως αυτά τα χρήματα πάνε από εκεί στις ε, Βρετανικές πρώην Μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, και ο Χουάνι από νησί προέρχεται. Επομένω γι' αυτό και τον καίει το θέμα. Δεν ξέρω πόσο ο Βρετανό το θέλει να απαντήσει. Βεβαίω. Σε αυτό το πρώτο ερώτημα. Γι' αυτό και δεσμευτικά πρότυπα ο Ολλανδό συνάδελφο τα είπε στο κείμενο του στο τι προβλέπει να γίνεται με αυτές τις ε, εκτίσει που ίσως πιο αποτελεσματικά μπορούν να καλυφθούν, υπάρχει μεγαλύτερη υποπτία την Ένωση επ' αυτών. Δεν συμφωνώ 100% μαζί του. Και να, κοιτάξτε τι έγινε με τα νησιά Κέιμα και τι νομολόγησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. όσον αφορά με την οδηγία τη αποτανίευση, για το αν μπορεί να ισχύσει στα νησιά Κέιμαν, δεν ξέρω, ίσω ο ίδιος ο Ρωσλανδός συνάδελφο διαφωνεί, αλλά επίσης διαφωνώ και με την ε, ιδέα ότι υπάρχει τώρα νομικό κενό. Σας είπα ποιες είναι οι αμφιβολίε προηγουμένω. Αλλά βέβαια θα να βασίλειο και αυτέ οι προεκκλήσει ότι ενεργούν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Δεν θέλουν διπλά πρότυπα. Και ότι και, να υπάρχει, να υπάρχουν δύο μέτρα στο από αυτού που του επικρίνουν. Νομίζω ότι όλες αυτές οι πρώην θέλουν ε, να μείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό δείχνει πώ βλέπουν τον ρόλο του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο ωφελούνται από αυτό και πόσο θέλουν να ακούγεται η φωνή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβούνται μήπω όλα αυτά χαθούν. Δεν βλέπουν τον Brexit σαν ευκαιρία να εκμεταλλευτούν την ναι, αυτή η ελευθερία τους. Έτσι να παρακάψουν τους κανονισμούς και την εποπτεία. η ΙΠΑ, ο ΩΣΑ και άλλοι συνεχίζουν να τους ασκούν πίεση. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό το κακό σενάριο θα υλοποιηθεί και θα έχουμε τέτοιου είδους ροές προς τις προεκτήσει αυτές. Δεν θέλουν να δίνουν αυτή την εικόνα. Θέλουν να δίνουν την εικόνα κάποιου αξιόπιστου χρηματοοικονομικού διαχειριστή, ας πούμε, Καλά, δεν υπάρχουν και επιχειρήματα περί του αντιθέτου. Πάντω για το ρόλο τη Ένωση δίνω τη σκητάλη στον Ολλανδό συνάδελφο. Ευχαριστώ. Η κυβέρνηση του Βασιλείου δεν μπορεί να φέρει σε πέρα αυτό. Ίσως θα πρέπει να αξιοποιήσει τις εξουσίες ε, του Κοινοβουλίου και επειδή δεν έχει πολλά χρήματα με τις επιδοτήσεις ενδεχομένω από τις Βρυξέλλες ε, θα μπορούσε κάτι να γίνει. Νομίζω ότι όλοι το ίδιο πράγμα έχουμε βιώσει. Υπάρχει και το προήμιο σε αυτή τη συμφωνία για την υπερποντέδα και μιλάει και για τη διαφάνεια που είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο για τη χορήγηση των επιδοτήσεων. Θα μπορούσα να μη χορηγούνται ή να επιστρέφονται αυτές οι επιδοτήσεις αν δεν πληρείται, πληρείται αυτός ο όρος της διαφάνειας και αν υπάρχουν προβλήματα και ανεπάρκειες. Είναι μια δυνατότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να περιορίσει και να αναστείλει τις επιδοτήσεις. Έχει τη διακριτική ευχέρεια. Καλό είναι λοιπόν να υπάρχουν και αυτή τη δυνατότητα χρήση πιο σκληρών μέτρων. Ο πρόεδρος αν δεν κάνουν πουλάκια τα μάτια μου, θα έλεγα ότι δεν εκπροσωπείται η ομάδα ECR, ούτε και η Άλντε. ενώ ότι δεν έχει βουλευτές εδώ. Το προσωπικό είναι πάντα εδώ, αλλά οι βουλευτές δεν είναι εδώ. Δεν κάνω λάθος, κάνω όχι. Επομένως, επόμενος ομιλητή είμαι εγώ, ο ίδιος, εκ μέρου τη Γκουε. Καταπληκτικά. Και το πρώτο μου ερώτημα θα ήταν το εξής. Μια από τις μελέτες λέει ότι απλώς έλεγχος της ροής ε, των χρημάτων που επενδύεται στις περπότες χώρες και δάφη σημαίνει απλά ότι μετατοπίζουμε όλο το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό αφορούσε κάποιους φόρους ως ποινή, κύρος κτλ. Πώς φτάσατε σε αυτό το συμπέρασμα είναι η πρώτη με ερώτηση. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, σε ένα έγγραφο του Foreign Office, λευκή βίβλος από τον Ιούνιο του 12 συγκεκριμένα, εκεί λέγεται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Κοινοβούλιο, έχει περιόριστη εξουσία να νομοθετεί για τα εδάφη, αλλά υπήρξε μια απόφαση το 2009 μόνο ε, για τα νησιά Τέρξ και Κάικος όπου υπήρξε κάποια παρέμβαση. Δηλαδή, ουσιαστικά, ενώ έχει αυτή τι εξουσίε στο Ηνωμένου Βασίλειο, επιλέγει να μην τι ασκεί. Υπάρχει εδώ κάποιο συνταγματικό πρόβλημα ή όχι. Ή είναι ένα θέμα που είπατε και πριν, ότι δηλαδή είναι επιφυλακτική και απρόθυμη για να μην χάσουν την οικονομική αυτάρκεια. Και τέλος, αν δούμε και τις τρεις μελέτες, Νομίζω ότι και η Γρυλανδία ε, αναφέρεται και τα γαλλικά υπερπαντή εδάφη. Ε, μπορεί να μην ήταν ποτέ σε κάποιο κατάλογο φορολογικών παραδείσων. Μπήκαν όμως. Τι γίνεται όμως με τα βρετανικά να εδάφη ακριβώς. Ε, ποια επιλογή, η επιλογή αυτή που έγινε, πού βασίστηκε και από τους τρεις σας. και στα παραρτήματα διαφέρουν τα ίντεξ. Είναι ένα πρόβλημα αυτός προς τη συγκρισιμότητα. Μπορείτε να δώσετε κάποια συνέχεια ενδεχομένω σε αυτό, μπορείτε να μας δώσετε κάποια εξήγηση. Ίσως μπορώ να απαντήσω το πρώτο ερώτημα, να απευθύνεται μέσα σε μένα, από την κατάλαβα. Θεωρητικά, η κυβέρνηση μπορεί μέσω εντολών να διαταγμάτων να ε, νομοθετήσει και να παρέμβει. Ουσιαστικά είναι η εξουσία της μοναρχίας και δεν χρειάζεται να περάσουν τα θέματα από την κοινοβουλευτική συζήτηση, να πάρουν κοινοβουλευτική έγκριση. Είναι ένας παλιός κοινοβουλευτικός μηχανισμός που χρησιμοποιεί όποτε ε, το χρειάζεται το Ηνωμένο Βασίλειο για το Σύνταγμα και για την νομοθεσία. Και όπως λέτε σωστά επιλέγει να μην ε, παρέμβει, είναι πολύ απρόθυμο το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως ε, ε, δώσατε εσείς ένα παράδειγμα, το παράδειγμα Τέρξ και Κάικος, ήταν κατά της τα εδάφη ήταν ένα πιο μακρινό παράδειγμα από ποινικοποίηση του σεξ μεταξύ ομοφύλων και Βλέπετε λοιπόν ότι πολύ σπάνια παρεμβαίνει το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν ανέκτησαν άμεσο έλεγχο στα νησιά Τέρφ και Κάικο, στο επίπεδο ε, κριτικής ήταν τεράστιο και από τη ΣΕΑ και από την Καραϊβική είχαμε αντίστοιχες αντιδράσεις. Επομένως, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένων για το κατά πόσο θα χρησιμοποιήσει την πυρηνική, αν επιτρέπει όρος αυτή, επιλογή και δεν το κάνει συχνά. Να πω κάτι για τη μεθοδολογία που επιλέξαμε. Αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στις τρεις πιο περίπλοκες περιπτώσεις. Γι' αυτό και δεν συζητήσαμε την περίπτωση και γιατί δεν είναι ιδιαίτερα προβληματική. Σε ό,τι αφορά το πώς θα εξελισσόταν η μελέτη, δώσαμε ευρία εντολή στους εμπειρογνώμονες, διότι από την αρχική έρευνα που κάναμε εσωτερικά, διαπιστώσαμε ότι ήταν διαφορετικά τα συστήματα και περίπλοκα και θελήσαμε να τους δώσουμε την ελευθερία να αναδυφίσουν στην περιπλοκότητα, η οποία μου φαίνεται ότι φάνηκε και ώρα από τις παρουσιάσεις τους. Και κάναμε αυτή τη συνολική εισαγωγή προσπαθούμε να συγκρίνουμε εσωτερικά τις τρεις μελέτες σε διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή νομικό πλαίσιο, οικονομικό και πολιτική επιρροή που έχει η χώρα μέλος στα υπερπόντια εδάφη της, προσπαθώντας να τα βάλουμε σε μια οπτική συγκρισιμότητα σε αυτά τα τρία. Σας ευχαριστώ πολύ και επειδή δεν θέλω να φανώ άδικος, και να δώσω στον εαυτό μου περισσότερο χρόνο από ό,τι έδωσα στους άλλους. Πολύ σύντομα, αν μπορεί κάποιος εκ των ομιλητών να εξηγήσει αν βλέπετε κάποια δυνατότητα φορολόγηση στην πηγή ε, των ε, ε, διακινουμένων ποσών ώστε να διευκολυνθεί η κατάσταση εκεί. Αν είναι δυνατόν σε ναι. μισό λεπτό. για τις γαλλικές υπερπόντιες κτήσεις υπάρχουν κάποιες κρατήσεις στις πηγές και κάποιες κυρώσεις που προβλέπονται και οι οποίες επιβάλλονται για παράδειγμα σε επιστοτικά ιδρύματα όταν οι ε, κρατήσεις στην πηγή δεν γίνονται ορθά για τα εισοδήματα όπου μπορεί αυτό να γίνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, και μια επιχείρηση είναι πολύ πιο δύσκολο παρά ο τόκο που πληρώνεται από μια επιχείρηση. Από μια τράπεζα, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ. Ο επόμενος είναι κάποιος από τους πρασίνους που δεν βλέπω όμω κανένα εδώ παρόντα. EFDD. David Cobbett. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κλέγγ, στις ε, χώρες αυτές περιοχές δεν είναι είναι όλοι τόσο δυστυχισμένοι από τον Brexit. Δεν θέλουν την, ε, τον ανακατεύτο Βασίλειο. Ο, ε, δεν το θέλουν. Και είχαμε εμπορική συμφωνία δεκαετία του 70 και μας ξεγέλασαν οι κυβερνήτες. Δεν είχαμε να μπούμε έτσι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με σημαία, εθνικό ύμνο, κυβέρνηση και όλα τα άλλα του πακέτου. Γιατί θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακατευτεί σε αυτές τις πρώην Δεν έχει καμία δουλειά. Εμείς πάμε για Brexit και αυτό ψήφισε ο Βρετανικός λαός. Το πρόβλημα βέβαια πάντοτε ποιο είναι. Το θέμα το, το φορολογικό. Και έχουμε αυτούς τους γραφειοκράτες με τις μισθάρες τους και τις φοβέρε τους συντάξεις. Μεγάλα είναι τα προβλήματα που δημιούργησε το καταρρεύσαν ευρώ. Είδα τι έγινε στην Νότια Ευρώπη. Το ευρώ έχει μόνο πολιτική στήριξη, καμία οικονομική ε, ουσία. Μα είναι δυνατόν να μας ε, ε τι θα κάνουμε στη χώρα μας ή στις πρώην κτήσεις, γιατί εσείς τα καταφέρατε. Πάμε να μην ανακατευτούμε, δεν ανακατευόμαστε σε αυτές τις επικράτειες. Θέλουμε να είναι ανταγωνιστικέ και, και όσον αφορά τα φορολογικά και βέβαια να μην ε, υπάρχει έγκλημα. Οπότε αν δεν υπάρχει έγκλημα δεν ανακατεύουμε. Εμεί αυτό ονομάζουμε δημοκρατία. Δεν ξέρω Μήπω θα πρέπει να αντιλήσει από αυτήν την αντίληψη για δημοκρατία συμπράζουν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ανακατευόμαστε ούτε στα εσωτερικά του να ανακατεύουμε στα δικά μα εσωτερικά, ούτε στο τι γίνεται σε αυτές τις κτίσεις. Ας φροντίσει η κυβέρνησή τους. Θα ήθελε κάποιος να απαντήσει η Βασίλισσα ή κάποιος άλλος, ο καθηγητής Κλέγκ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Αυτές οι προεκτήσεις προβληματίζονται για τις επιπτώσεις του Brexit όσον αφορά την ελευθερία διακίνηση, όσον αφορά την πρόσβαση στην ενιαία αγορά, όσον αφορά τους πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση που βοηθούν την οικονομική τους ανάπτυξη. Είδατε τι έγινε και με την ψήφο του Γιβραλτά. Δεν θέλουν να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτούς τους λόγους. Καλά, είναι και τα θέματα τα εξωχώρια, τα οικονομικά. Γίνανε και κάποιες ε, εκθέσεις και μελέτες για να δουν τι θα γίνει με τις επιπτώσεις του δημοψηφίσματος, αν φύγει δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση από την Ένωση. Ε, να δούμε τα επόμενα χρόνια τι θα βγει. Μπορώ να δευτερολογήσω. Ναι, ναι, ναι. Ε, είδατε τι με το, με το Γιβραλτάρ που αναφέρετε. Θα ήταν πολύ χειρότερα αν ήταν στην Ισπανία δημοσιονομικά. Είδατε τρομερή ανεργία που έχει η Ισπανία και όλο το, το εμπορικό ατού του Γιβραλτάρ, αν ε, πάει στην Κώστα Ντελσόλα, αντίο αυτό το εμπορικό πλεονέκτημα. Το ίδιο και με την υπόλοιπη χώρα. Τι πρόβλημα θα πάνω σα λέω κύριε, το θέμα δεν είναι ότι βοηθά την ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πληρώνει ο βρετανό φορολογούμενο και ο Γερμανό φορολογούμενο. Δεν έχει λεφτά να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει χρεοκοπήσει. Τα δίνει το, η Βρετανία μέσω τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύτερα να αφήσετε στην ησυχία του τι προεναπικίε μα. Έχω μια ταπεινή πρόταση, λέει ο πρόεδρο, γιατί έχουμε αυτό το συγκρότημα, το έτσι που έλεγε Don't look back in anger. Μεγάλη σου επιτυχία. Είναι γεγονό το Brexit και θα το χειριστούμε. Νομίζω ότι εσεί κύριε Κόμπερν και εσεί πληρώνεστε από του Βρετανού φορολογούμενου. Άρα α το αφήσουμε. Εκτό μικροφώνου κύριο Κόμπερν. Ναι, ναι, ναι, και εγώ, και εγώ, έχετε δίκιο. Εκτός μικροφόνο παρατήρηση του κ. Κόμπερ. A very short comment by Κύριο μια στην παρατήρηση και προχωρούμε. Κλέγγ, δυστυχώς. Για όλα αυτά δεν υπάρχει μαύρο και άσπρο όπως είπατε ή χαμένο ή κερδισμένο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει διαβήματα στην κυβέρνηση. Ότι δηλαδή όλοι αυτοί οι πόροι που θα χαθούν από το Brexit ε, ή μάλλον όλα αυτά τα οποία, τα οποία έχετε ισχυριστεί ότι πηγαίνουν στις αυτές τις, ε, τις περιοχές δεν έχουν πραγματικά εκταμιευτεί. Κύριο Κόμπερν απαντά εκτός Θα τις φρόντιζε αυτές τις περιοχές πολύ καλύτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όχι να τα δίνουμε στη μαύρη τρύπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παίρνουν ε, πέντε ροδεκάρες τελικά αυτές οι κτίσεις. Πάντα φταίει ο ενδιάμεσος, ο πρόεδρος. Ολοκληρώθηκε αυτό το θέμα. Και τώρα, η ΕΝΕΦ δεν έχει κάποιον αγορητή στην αίθουσα, άρα... Ο τελευταίος είναι ο κύριος Ροζάτη. Σας είναι το λόγο, αλλά δεν τον θέλατε. Σας εξέπληξε εκτός μικροφώνου ο κύριος Ροζάτη. Η μεγαλύτερη έκπληξη για σήμερα είναι ότι τα καταφέραμε να τηρήσουμε τα χρονικά πλαίσια της συνάντησης. Οπότε να ευχαριστήσω τους ερευνητές μας που ήρθαν για να συζητήσουμε, άρα και που ήρθαν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Και τώρα, οι συνεισηγητές. Ας ολοκληρώσουν, αλλά δεν είναι εδώ. Οπότε, ο ίδιος θα ευχαριστήσω όσους ήρθαν εδώ. Αλλά και τους διερμηνείς που θα έπρεπε όλα σε να τα μεταφράσουν. Και πολλέ φορέ τα είπαμε πολύ γρήγορα και επίση να ευχαριστήσω και του συνεργάτε μα και τι πολιτικέ ομάδε που έδειξαν την υπομονή να μείνουν μαζί μα σήμερα. Δεν έχουμε για τα διάφορα κάτι άλλο και η επόμενη συνάντηση θα είναι στι 4 Πέμπτου του Εναστότο έτου 9 με 12.30 εδώ στι Βρυξέλλε. και σα ευχαριστώ. Καλό βράδυ. New round of applause for the British taxpayer, eh? And <laughs> who pays my bill.